Dear colleagues, I would like to start the meeting. I hope everything is clear and we can start the meeting. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Με το σημείο 1 της μερίσιας διάταξης. Έγκριση της μερίσιας διάταξης. είναι τελικά παράδοση τελευταία στιγμή να, να υποβάλλονται αιτήματα τροποποίηση. Ο Πάλο Ράντζο, που είναι συγκεκριτή για την εφαρμογή των συνθήκων, τη συνθήκη που αφορούν τα εθνικά κοινοβούλια, το προβλέπουμε για το απόγευμα 5.45 με 6 και 10. Θα γίνει αντιστροφή με τον Νταν Πρέντα ο Παύλο Ράντζελ θα παρουσιάσει το θέμα του 10 και 30 με 10 Ο Παύλο Ράντζελ θα παρουσιάσει το θέμα του. Το δεύτερο είναι το αίτημα του εισηγητή γνωμοδότησης Πασκάλ Ντιουάν Υποτίθεται ότι πρέπει να προτείνουμε το ρόλο, τον ε, γνώμη στο τζούρι για τους κανόνες, για τις γενικές αρχές που αφορούν τους μηχανισμού για τον έλεγχο των κρατών μελών από την Κομισιόν για την ε, άσκηση των, ε, τον έλεγχο των κρατών μελών στην Κομισιόν για την εφαρμογή των εφαρμοστικών αρμοδιοτήτων, αλλά επειδή χρειάζεται να, να συνεχιστούν οι συζητήσεις θα το αφαιρέσουμε από τη μέσα διάταξη και τώρα προτείνεται και άλλη μια αλλαγή, θα γίνει ένα αλλαγή μεταξύ του σημείου του Γκέργη Τσιόπλιν για, τις ευρωπαϊκές, για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών με την έκθεση για τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα ακούσουμε πρώτα τον Γκέργη Τσιόπλιν για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία των Πολιτών, το ECI. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσει, ε, μπορούμε να περάσουμε στο σημείο 2 τη ημερήσια διάταξη, που είναι ανακοινώσει τη Προέδρου. Εδώ θα ήθελα να σε ενημερώσω ότι Υπάρχει ένα θέμα που ορισμένοι μπορεί να το έχετε ξεχάσει. Υπάρχει μια ομάδα εργασία που δημιουργήθηκε μετά την διοργανική συμφωνία για την καλύτερη νομοθέτηση, για είναι μια ομάδα εργασία για την εφαρμογή και ερμηνεία της διοργανικής συμφωνίας για την καλύτερη νομοθέτηση. Η ομάδα αυτή έχει συναντηθεί 8 φορές και μαζί με την Τζούρι ε, εξετάσαμε όλα τα κεφάλαια της διοργανικής συμφωνίας. Είχαμε και ακροάσεις. με τους ειδήμονες για τα θέματα αυτά. Επίσης κάποιοι συνάδελφοι συμμετέχουν σε διαπραγματεύσεις για την διοργανική αυτή συμφωνία για δύο θέματα. Το πρώτο θέμα αφορούν, αφορά τους ε, Μπροκ και Μπέρντ Λάγκε και συζητούν το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τις διοργανικές ε, σχέσεις στα πλαίσια των διεθνών συμφωνιών. Συζητούν κάποια πρακτικά θέματα, κάποιες πρακτικές διευθετήσεις και για το θέμα αυτό. Και επίσης, ο κύριος Σάιρ της Τζουρί και ο από πλευράς μας. Διαπραγματεύονται λοιπόν για τα κριτήρια για την εφαρμογή των κατεξιοδότηση και εφαρμοστικών πράξεων. Η ομάδα αυτή έχει αναπτύξει έντονη δραστηριότητα και μετά τις διακοπές θα σας ενημερώσουμε για το πότε πρέπει να αναμένεται η τελική έκθεση από τον Ρίτσαρτ Κόρμπετ. Σχετίζεται με το πώς θα καταλήξουν οι εργασίες αυτής της ομάδας εργασίας. Να περάσω τώρα στο 3. Έγκριση των πρακτικών των συναντήσεων μας. Έχουμε συγκεκριμένα τη συνάντηση της 9ης Φεβρουαρίου. Τώρα τον Ιούλιο. άργησε μετάφραση. Ωραία. Τα έχετε και θα κρυθούν αν δεν ε, υπάρξουν αντιρρήσεις μέχρι το τέλος της συνεδρίασης. Τώρα, να περάσουμε στο σημείο 5 της ημέρης διάταξης αναθεώρηση του κανονισμού για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία των Πολιτών. Το έχουμε συζητήσει ήδη επανειλημμένα. Ε, ε Γιώργη, ε, Σόπφλιν, έχεις τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ και καλημέρα Όσοι παρακολουθούν αυτή την ιστορία γνωρίζουν το θέμα αυτό το συζητάμε πολύ καιρό. Από την προηγούμενη ήδη θητεία. Το άρθρο 11 της συνθήκης δίδει τη δυνατότητα σε ένα εκατομμύριο πολιτών εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου από έναν αριθμό χωρών να αναλάβουν πρωτοβουλία για να υπάρξει κάποια τροποποίηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας μέσω υποβολής πρότασης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα εξαρτάται από το πώς τις υπολογίζουμε, αλλά έχουν υπάρξει 60 τροπολογίες. Αλλά με μία μερική εξαίρεση καμία δεν έχει καταλήξει σε νομοθετική δράση. Αυτή ήταν ε, η κατάληξη της προηγούμενης εκθεσής μου και άρα δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι τα πάει και τόσο καλά ως δυνατότητα. Αλλά είναι το ιδανικό όργανο για να βοηθήσει την προσέγγιση των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και να τονίσω επίσης ότι αξιοποιείται ήδη σε δύο κράτη-μέλη, Φιλανδία και Λετωνία, και από ό,τι καταλαβαίνω με επιτυχία, αλλά δεν έχω στοιχεία. Πολύ θα ήθελα όμως να μου αποσταλούν. Ένα βασικό θέμα που είναι και πολιτικής και νομικής φύσης είναι ότι το άρθρο 11 λέει «Καλή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα το θέμα είναι τι σημαίνει καλή. Αν είναι απλώ μια πρόσκληση προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να πει ευχαριστώ για την πρόσκληση, θα σα πούμε τι θα γίνει. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Τώρα κοίταξα πώ μεταφράζεται σε διάφορε γλώσσε, αυτέ που γνωρίζω, και είναι απόλυτα σαφέ. Είναι μια λέξη του στυλ ε, invité, invitar, και στα ουγγρικά είναι ακόμη πιο αδύναμη η λέξη που χρησιμοποιείται. Δηλαδή τι εννοώ, δεν επιβάλλεται υποχρέωση στην Επιτροπή να αναλάβει κάποια πρωτοβουλία εάν υπάρξει αυτό το εκατομμύριο υπογραφών σε ένα χρόνο, εάν υπάρχουν λοιπόν όλες οι προϋποθέσεις. και αν από νομική άποψη ε, μπορεί να γίνει αποδεκτό το αίτημα. Σε αυτή την ε, κατάσταση είμαστε τώρα. Η στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ποικίλει. Όταν υπέβαλα την ε, προηγούμενη έκθεση ήταν πολύ φιλικές συζητήσεις και είχα την εντύπωση ότι ήταν διατεθειμένοι να δεχθούν κάποιες τροποποίησεις, μάλλον να προτείνουν κάποιες τροποποιήσεις είναι ο κανονισμός 2011 είναι ο κανονισμός που υποτίθεται ότι ε, ρυθμίζει πώς θα ασκεί την πρωτοβουλία αλλά μετά δεν παρουσιάστηκε στο πρόγραμμα εργασίας της Κομισιόν και στα πρακτικά κάποια συνάντηση των επιτρόπων η πρωτοβουλία αυτή περιγράφηκε ως επικίνδυνη. Τώρα αυτά είναι πολύ ακραία να θεωρούν επικίνδυνη μια δυνατότητα προσέγγισης της, ε, των πολιτών προς την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι είναι κάπως ε, ιδιόρυθμη προσέγγιση για το τι είναι δημοκρατία. Νωρίτερα φέτος υπήρξε και η μερίδα για το ECI, όπου συμμετείχε και ο αντιπρόεδρος Τίμερμανς, ο οποίος ξαφνικά ανήγγειλε ότι είναι καταπληκτική δυνατότητα το ECI και θα κάνει μια δημοσιακή βούλευση η οποία νομίζω λύγει στις 16 Αυγούστου, οπότε δεν ξέρουμε τα αποτελέσματα μέχρι τώρα. Μεταστράφει λοιπόν η άποψη της Κομισιόν και ίσως αυτό εν μέρη να σχετίζεται με, το αυτό με αυτά που κάνουμε εμείς εδώ, αλλά ίσως να κάνει περισσότερο και με τις δύο υποθέσεις που πήγαν στο δικαστήριο και τις οποίες έχασε στην ουσία η Κομισιόν για το τι είναι αποδεκτό και τι όχι. Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα. Η Κομισιόν τώρα μοιάζει διατεθειμένη, αν αυτό σημαίνει ότι θα μας υποβάλει πρόταση αναθεώρησης του κανονισμού αυτού, θα το δούμε και τι τροπολογίε θα μας προτείνει, τι τροποποίηση. Αυτά λοιπόν και προσβλέπω και στη δική σας συμβολή. Ελπίζουμε λοιπόν να Υποβάλλουμε μία έκθεση νομοθετικής πρωτοβουλίας που τις προσέχει περισσότερο η Κομισιόν, ούτως ώστε να γίνει πιο εύχριστο το μέσο αυτό, γιατί είναι κάπως δύσχριστο, όπως για παράδειγμα, πώς παρουσιάζεις τον εαυτό σου. Υπάρχουν 28 διαφορετικά συστήματα και βεβαίως ε, ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν υπάρχουν ταυτότητες, άρα πώς ε, επιβεβαιώνεται η ταυτότητα των υπογραφών Στην Ουγγαρία λέγεται ότι πρέπει να δώσεις και το γένος της μητέρας σου. Δεν ξέρω γιατί τώρα, ίσως είναι απομεινάρι της Αυστρο-Ουγγαρίας. Είναι εντελώς παράλογο, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Πολλές προτάσεις στο κείμενό μου θέλουν να κάνουν πιο εύχριστο το μέσο αυτό, αυτή τη δυνατότητα. Και θα ήθελα το Κοινοβούλιο να παίξει ενεργό ρόλο στη διαδικασία αυτή και αν κάποια πρωτοβουλία καταφέρει να συγκεντρώσει ένα εκατομμύριο υπογραφών, τότε λέω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να συζητήσει τις πρωτοβουλίες των πολιών που επιτυχώς ε, πληρούν όλα τα κριτήρια που, που καθορίζει ο κανονισμός. Και οι συζητήσεις μπορούν να καταλήξουν με την υιοθέτηση, με την έγκριση πρότασης ψηφίσματος. Δηλαδή, θεωρώ ότι εάν συγκεντρωθεί ένα εκατομμύριο υπογραφών, το Κοινοβούλιο πρέπει να κάνει γνωστή αυτή την πρωτοβουλία για να υπερβούμε αντιστάσεις στην ε, υιοθέτηση νομοθετημάτων όπως ζητούν οι πρωτοβουλίες. Τέλος, συζήτησα σε σημαντικό βαθμό με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών συζήτησα για το αν είναι άμεση δημοκρατία αυτή η πρωτοβουλία ή όχι. Τώρα είναι τεχνικής φύσης. Εγώ θεωρώ ότι βεβαίω δεν είναι σαφώς αντιπροσωπευτική δημοκρατία αλλά ούτε άμεση δημοκρατία. Είναι sui generis. Που σημαίνει πως δεν ξέρω πού να ταξινομήσω αυτή την δυνατότητα. Και αυτό είναι. Δεν νομίζω ότι είναι παραχώρηση στο λαϊκισμό. Υπάρχουν αρκετές ασφαλιστικές δικλίδες, ούτως ώστε να έχουμε υπεύθυνη δράση από πλευρά τη κοινωνία των πολιτών και στι συζητήσει που κάναμε στην προηγούμενη θητεία, ορισμένοι ανησυχούσαν ότι είχαμε διάφορε γελίε πρωτοβουλίες ή ενδεχομένως και κακόβουλες. Αλλά δεν συνέβη, το αντίθετο συνέβη. Νομίζω ότι υπήρξαν μια σειρά από πολύ υπεύθυνε προσπάθειες για να ασχοληθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άρα το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλέγμα με σοβαρά θέματα, αλλά δεν κατέληξαν μέχρι στιγμής. Και κάτι άλλο που δεν ε, το συμπεριέλαβα στην προηγούμενη έκθεση, αλλά νομίζω ότι πρέπει να είναι ένας στόχος. Πρέπει να υπάρξει μια ευρωπαϊκή ψηφιακή δυνατότητα ταυτοποίησης των πολιτών. Νομίζω ότι είναι τμήμα της ψηφιακής, ε, του ψηφιακού θεματολογίου που συζητάει το Κοινοβούλιο και θα διευκόλυνε την συλλογή υπογραφών, για παράδειγμα και θα διευκόλυνε και την ενημέρωση για αυτές τις δραστηριότητες. Αυτά σε γενικές γραμμές και ελπίζω ότι θα είναι συναρπαστική και δική σας συμβολή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Τζορτζ. Θα ήθελα να ρωτήσω καταρχήν οι ανισχυώδεις θα ήθελα να λάβουν το λόγο. Σιλβί, είσαι εδώ. Ωραία, η κυρία Κάφουμα, λοιπόν. Ευχαριστώ να ζητήσω συγγνώμη από τον εισηγητή. Ήμουν στην Επιτροπή Τζούρι για τη συζήτηση με την Εστονική Προεδρία. Δεν ήξερα ότι τώρα θα τροποποιηθεί η μερίσια διάταξη και θα αντιστραφούν αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή. Περιέλαβε πολλά σημαντικά θέματα. Εδώ και πολύ καιρό έχουμε μια ιδιαίτερα έντονη συζήτηση για την τροποποίηση του κανονισμού αυτού και χαίρομαι που με ελάχιστες εξαιρέσεις συμφωνούμε για τα ε, θέματα αυτά και τα βλέπω στην έκθεσή του. Να αναφέρω ορισμένα θέματα που θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικά. Υπάρχουν προτάσεις για τις οποίες πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε, ούτω ώστε για να τις εφαρμόσει η Κομισιόν, δηλαδή να υποβάλει νομοθετικές προτάσεις μέχρι τέλους του χρόνου. Τι είναι πολύ σημαντικό. Το θέμα της ε, μερικής καταχώρησης μιας τέτοιας πρωτοβουλίας, αυτό σχετίζεται και με την ε, απόφαση του δικαστηρίου. Η προθεσμία για την ε, συγκέντρωση υπογραφών είναι πολύ σημαντικό. Εγώ θα ήθελα αυτός ο αυτοματισμός μεταξύ της έναρξης των υπογραφών και της καταχώρησης να αρθεί. Οι οργανωτές να έχουν τη δυνατότητα να καθορίζουν οι ίδιοι πότε ξεκινάει η συλλογή υπογραφών. Αυτό το περιέλαβε ο όπως και το θέμα της εναρμόνισης και απλούστευσης της διαδικασίας συλλογής υπογραφών. Ναι, υπάρχει δυνατότητα να συμμετέχουν στη συλλογή υπογραφών στη χώρα διαμονής και το θέμα της ευθύνης των διοργανωτών είναι σημαντικό ότι έχουν ευθύνη μόνο για ενέργειες ε, που παραβαίνουν τον νόμο. Κάτι άλλο, αν ε, δεν γίνει δεκτή μία καταχώρηση από την υπογραφή, η Κομισιόν να είναι υποχρεωμένη να δώσει μία αναλυτική και κατανοητή αιτιολόγηση. Υπάρχει μία πρόταση στην έκθεση που τη στηρίζω ιδιαίτερα, ότι όταν υπάρχουν επιτυχημένες τέτοιες πρωτοβουλίες, ο εισηγητής προτείνει πέρα από την ε, ακρόαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να γίνεται και συζήτηση στην Ολομέλεια για αυτές τις επιτυχημένες πρωτοβουλίες των πολιτών. Και ενδεχομένως, mail λέει στα αγγλικά, ενδεχομένως λοιπόν, να ε, εγκρίνεται και ψήφισμα. Νομίζω πως ε, είναι πολύ καλή πρόταση. Έτσι όλοι οι πολίτες οι οποίοι έχουν ε, υπογράψει θα καταλαβαίνουν, θα αντιληφθούν πόσο σοβαρά παίρνουμε υπόψη το αίτημά τους. Σοβαρή βελτίωση. Τώρα να πω λίγα λόγια για τα σημεία όπου θεωρώ ότι ίσως πρέπει να γίνει περαιτέρω συζήτηση. Θέματα που δεν βλέπω δηλαδή. Θέλω να αφαιρθώ σε αρκετά θέματα. Πρώτον, θα πρέπει να δούμε περαιτέρω εάν θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να υποστηριχθεί και οικονομικά μια τέτοια πρωτοβουλία. Για παράδειγμα, μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων όπως η Ευρώπη για τους πολίτες ή ισότητα δικαιωμάτων και ενωσιακή ηθαγένεια, όχι βέβαια με μεγάλα ποσά, αλλά μια μικρή οικονομική στήριξη θα μπορούσε να βοηθήσει τις πρωτοβουλίες αυτές εφόσον ε, ξεκινάνε να καταλήγουν κιόλα. Κάτι άλλο βασικό το γνωρίζει και ο συνάδελφος Σέπφλιν από τις συζητήσεις που κάναμε και πριν από δύο χρόνια. Είναι το θέμα της ελάχιστης ηλικία για την υπογραφή. Όπως ξέρουν οι συνάδελφοι, υπάρχει ένας παραλογισμός. Αν το συνδέσουμε με το ενεργό δικαίωμα συμμετοχής σε εκλογές, οι πολίτες της Αυστρίας μπορούν από τα 16 να συμμετέχουν, σε όλες τις άλλες χώρες όχι. Θα πρέπει να το δούμε αυτό το θέμα. Γιατί να συνδέεται με το ενεργό δικαίωμα συμμετοχή στι εκλογέ, στι ευρωεκλογέ. Γιατί πρέπει να είναι προπόθεση. Πρέπει να υπάρξει ενιαία ρύθμιση στην Ένωση για την ελάχιστη ηλικία και να είναι 16, να προτείνουμε 16 νομίζω πως θα ήταν ε, ένα σημαντικό μήνυμα της εμπιστοσύνης που έχουμε προς τους νέους, προς τη νέα γενιά, που νομίζω ότι με πολύ υπεύθυνο τρόπο θα υπέγραφε τέτοιες πρωτοβουλίες. Θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στη διαμόρφωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να συμμετάσχουν, να συμμετάσχουν ενεργά. Κάτι άλλο που δεν βλέπω. να μπορούν να υπογράφουν και άτομα με ειδικές ανάγκες. Και εδώ υπήρξαν διάφορες ε, γνωμοδοτήσεις. Είναι δύσκολο να υπογράψουν τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Πρέπει να το δούμε περαιτέρω. Τελευταίο. Που για μένα είναι σοβαρό θέμα και δημιουργεί δυσχέρειε. Προτείνει ο κύριο Σέπφλιν οι πρωτοβουλίες αυτές να μπορούν να παρεύουν στην ε, τροποποίηση μιας ε, υποεξέλιξη νομοθετικής διαδικασίας. Πώς θα εφαρμοστεί αυτό στην πράξη. Η Κομισιόν έχει κάνει μια νομοθετική πρόταση, εμείς ως Κοινοβούλιο τη συζητάμε, όπως και το Συμβούλιο, και τώρα έρχεται μια πρωτοβουλία των πολιτών και λέει κάτι, οτιδήποτε, ότι θα κάνει τότε τι θα πρέπει να κάνει η Κομισιόν, να αποσύρει την νομοθετική πρόταση. Δεν βλέπω πώς μπορεί να λειτουργήσει κάτι τέτοιο. Εφόσον είναι υποεξέλιξη. Δεν είναι δυνατόν να παρεμβαίνει σε μια τέτοια υποεξέλιξη νομοθετική διαδικασία, μια τέτοια πρωτοβουλία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι είναι γενικά πολύ καλή έκθεση και χαίρομαι ιδιαίτερα. Και προσβλέπω μάλιστα στην επικοδομητική συνεργασία, ελπίζοντας ότι θα βελτιώσουμε αυτό το μέσο, θα το κάνουμε πιο εύχριστο και ότι θα πρέπει να γίνει πραγματικά success story. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Ο κ. Γευτός και για την ECR θα σας παρακαλέσω βέβαια να περιοριστείτε στο χρόνο που έχουμε διαθέσιμο. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα κάνω ό,τι μπορώ. Ήθελα να ξεκινήσω κάνοντας μία αναφορά στις συστάσεις που μας παρουσιάζει ο κύριος Σέπφλιν για το, και το κατά πόσο θα μπορούσαν αυτές οι πρωτοβουλίες να γίνουν πιο ευέλικτες στην συλλογή υπογραφών, στην καταχώρηση αυτών και στη συνέχεια που θα δοθεί. Συμφωνώ δεν θα απευθύνουμε απλώς ένα κάλεσμα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά πρέπει να ορίσουμε τι είδους ορολογία θα χρησιμοποιήσουμε. Καταρχήν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οποιαδήποτε στιγμή απορρίπτει τέτοια πρωτοβουλία θα πρέπει να το τεκμηριώνει επαρκώς, γιατί εμείς δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με ε, το εξή σενάριο. Εμείς μένα ενθαρρύνουμε τους πολίτες να παρουσιάζουν τέτοιου είδους πρωτοβουλίες και κατόπιν αυτό, ε, σε αυτό να μην δίνεται συνέχεια, από ε, την ίδια την δράση των ευρωπαϊκών θεσμών, να μην δείχνουν το απαραίτητο ενδιαφέρον. Οπότε οι συστάσεις αυτές και το κομμάτι ε, που συμπεριλαμβάνει τη συζήτηση που θα έπρεπε να γίνεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πέραν των ακροάσεων είναι κομμάτια τα οποία εγώ σίγουρα μπορώ να δεχτώ. Τώρα, για τα όσα είπε η προηγούμενη ομιλήτρια, να σας πω πως ε, σέβομαι πάρα πολύ αυτά τα σχόλια για την χρηματοδότηση των πρωτοβουλειών των πολιτών ε, τη στιγμή που ξεκινάνε. Όμως, αυτό που πρέπει να ε, εξασφαλίσουμε είναι η αμεροληψία. Εμείς θα προσφέρουμε τη θεσμική στήριξη για αυτές τις πρωτοβουλίες. Ναι, αλλά δεν μπορούμε να προσφέρουμε χρηματοδότηση, γιατί διαφορετικά θα μας ε, κατηγορήσουν για έλλειψη αμεροληψίας. Τώρα, όταν αναφερόμαστε στον περιορισμό, τον χρονικό, δηλαδή την ηλικία πριν της οποίας δεν μπορεί κανείς να υπογράψει με τέτοιου είδους πρωτοβουλία. Δεν είμαι σίγουρος για το ποια είναι η κατάλληλη τακτική, θα το δούμε, γιατί θα πρέπει αυτό να αποτελέσει ένα πραγματικό ευέλικτο μεν, αλλά πολιτικό δικαίωμα. Δεν είναι εδώ Τον ε, υποκαθιστά κανεί, Γκούε, υπάρχει κανείς. Χέλμουτ, ως σκιώδης. Εκ μέρους της Μπάρμπαρα Σπινέλη θα μιλήσω, γιατί και η ίδια δεν μπορεί να παραστεί σήμερα και είναι σε άλλη συζήτηση, μου ζήτησε λοιπόν να σας μεταφέρω την άποψή της. Καταρχήν θα ήθελε να ευχαριστήσει τον εισηγητή για το σχέδιο έκθεσης και συμμερίζεται πολλές από τις απόψεις τις οποίες παρουσιάζει. Παράλληλα θα ήθελε να υπογραμμίσει πως είναι πεπισμένη πως ο μελλοντικός κανονισμός χρειάζεται πολιτική και όχι μόνο ε, τεχνική ε, τροποποίηση γιατί αυτή τη στιγμή είχαμε την απόφαση του ΔΕΚ για την TTIP και νομίζω ότι αυτό αποδεικνύει πως υπάρχει έντονος πολιτικός δισταγμός από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής να δεχτεί τέτοιου είδους πρωτοβουλίες. Αν θέλουμε ένα πιο ανοιχτό εργαλείο για τη συμμετοχική δημοκρατία, χρειάζεται να δούμε ποιες είναι οι, οι συνθήκες επί τις οποίες ένα τέτοιο αίτημα γίνεται αποδεκτό και επίσης τι ακριβώς σημαίνει νομικό μέσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά πόσο μπορούμε να αλλάξουμε τρέχουσα νομοθεσία μέσω αυτού του εργαλείου. Και στις 16 Ιουνίου ο κ. σε μια ακρόαση ακρόαση δήλωση πως λυπάται που η εμπειρία μας μέχρι σήμερα αποδεικνύει πως αυτές οι πρωτοβουλίες των πολιτών δεν ε, προχωρούσαν προς τα εμπρός το ευρωπαϊκό project γιατί συνήθως έχει να κάνει με θέματα επικαιρότητα πολύ φορτισμένα τα οποία ενδιαφέρουν περισσότερο τις μειοψηφίες παρά την πλειοψηφία των Ευρωπαίων πολιτών και γενικά οδηγούσαν στη δημιουργία ευρωσκεπτικιστικών ε, αισθημάτων. Νομίζει η κυρία συνάδελφος πως αυτό θα πρέπει να αμφισβητηθεί ως δήλωση και εμείς ως εκπρόσωποι των Ευρωπαίων θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε το σημείο αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα πρέπει να επιβάλλει κάποιες περιορισμούς που δεν ε, προβλέπονται από τον ε, κανονισμό, ε, από το άρθρο 11 των Ευρωπαϊκών ε, Συνθήκων, όπως επίσης και από το άρθρο 24 σχετικής νομοθεσίας. Γιατί δεν νομιμοποιούμαστε να αρνηθούμε την καταγραφή τέτοιου είδους πρωτοβουλίας των πολιτών με αυθαίρετο τρόπο και δεν μπορούμε αυθαίρετα να λέμε πως εκφράζουν μόνο τις απόψεις μιας μειοψηφίας ή πως δεν είναι δημοκρατικές. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να προχωρήσουμε σε τέτοιου είδους δράσεις οι οποίε δεν καλύπτουν τους στόχους μας που είναι να σεβαστούμε απόλυτα τα όσα προτείνουν οι συνθήκες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να έρχεται σε αντίθεση με την καταχώρηση των πολιτών γιατί για παράδειγμα, η το επιχείρημα που χρησιμοποίησε για την ε, TTIP ήταν πω δεν επρόκειτο για νομικό εργαλείο και νομική πρόταση το άνοιγμα των διαπραγματεύσεων, αλλά για τεχνικό μέτρο. Αυτό το επιχείρημα ξεκάθαρα δεν στέκει. Και νομίζω ότι το γενικότερο δικαίωμα των Ευρωπαίων πολιτών να συμμετέχουν στα δημοκρατικά τεκτενόμενα τη Ευρωπαϊκή Ένωση σημαίνει πως θα πρέπει παράλληλα να έχουν τη δυνατότητα να δράσουν όχι μόνο για να τροποποιήσουν το παράγωγο δίκαιο, αλλά παράλληλα για να μπορούν και να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή του σε κάθε είδου νομοθεσία και για τα τρία συγκεκριμένα άρθρα τα οποία ε, αναφέρει ε, ο εισηγητής, η συνάδελφος, στηρίζει το αίτημα των όσων παρουσιάζουν τέτοιου είδους ε, να προσφέρεται πρακτική καθοδήγηση, άρθρο 3, ε, πρακτική συνδρομή, άρθρο 3 και στο άρθρο 4, όπου αναφερόμαστε στο πρόβλημα που, στο οποίο στάθηκε και η κυρία Κάουφμαν, δηλαδή την τροπολογία τρέχουσας νομοθετικής πρότασης. Και η συνάδελφος προτείνει να δίνουμε τη δυνατότητα η πρωτοβουλία των πολιτών να προτείνει και νέες νομικές ε, πράξεις, κατάργηση υφιστάμενων και τροποποίηση ε, τρεχόντων, ε, τρεχουσών νομοθετικών προτάσεων. Τα λέει έτσι για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι και αναφέρεται στο 296 δεύτερη παράγραφο του, ε, της ε, συνθήκης. Και επίσης οι προϋποθέσεις για την συλλογή δηλώσεων στήριξης και εδώ χαιρετίζει την πρόταση του εισηγητή και λέει πως στο νέο κανονισμό θα πρέπει να παρουσιαστεί μια σύσταση προς τα κράτη-μέλη να έχουν μια ενιαία προσέγγιση για αυτές τις διαδικασίες. Άρα λοιπόν θα πρέπει οι υπογράφοντες να μπορούν να υπογράψουν ήδη από τη χώρα διαμονής αυτές τις πρωτοβουλίες πολιτών. Έχουμε ακόμα δύο συναδέλφους, η κυρία Τζέιμς και ο κύριος Χαουρέγγι. Θα σας δώσω, σας παρακαλώ το λόγο, αλλά να είστε σύντομοι αγαπητοί συνάδελφοι, δεν έχουμε χρόνο. Κανείς δεν μας λέει ποιοι είναι οι συγγητές. Σύντομα παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, θα... κοιτάξτε, έχει αντιστραφεί σειρά. Και δεν είναι διθέσιμο συνάδελφο, είμαι υποχρεωμένο να μιλήσω ονόματί του. Δεν είναι ότι θέλω να ενοχλήσω. Πάρα πολύ γρήγορα. Να αναφερθώ στα βασικά σημεία ε, που ο κ. Καμπά ε, θέλει να επιμείνει. Απλώ θέλω να τα παραθέσω, θα επιμείνω. Το πρώτο πράγμα που θέλει να αναφέρει, θέλει να ευχαριστήσει τον Ζορ για τη δουλειά που έκανε και πολύ γρήγορα θα διατρέξω αυτά που είπε η κυρία Κάφμαν. Υποστηρίζουμε το θέμα του ψηφίσματο του Κοινοβούλιο το, το Κοινοβούλιο να μπορεί τελικά να διασυνδεθεί με αυτή την κίνηση και να κάνει ψηφίσματα για κάποια κείμενα, ώστε να υποστηρίξει την προσέγγιση. Αυτό είναι σημαντικό. Τώρα για την ηλικία, στα 16 χρόνια. Εφόσον υπάρχει το δικαστήριο που, θα, που έχει τοποθετηθεί, οι πρωτοβουλίες όσον αφορά τη, τη Σύμβαση ε, Διεθνών Συμφωνών ο κ. Στέλι Καμπράς θέλει επίση ε, ενδεχομένω να επιτρέψουμε ε, τις, αυτές τις πρωτοβουλίες ε, για τις τροπολογίες των συνθήκων. Για τα υπόλοιπα, όπως το πείτε πάρα πολύ γρήγορα, προσπαθούμε να έχουμε διαφάνεια και ο κύριος ε, Τίμερμανς θέλει να και στην αρχή και στο τέλος να υπάρχει μια παρακίνηση όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν γίνονται οι και η δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν όλες οι επίσημες ε, γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για να μην ε, υπάρχει άλλου είδους επιλογή. Δεν μπορούσα να είμαι πιο γρήγορος, κυρία Πρόεδρε. Η κυρία Νταϊάν Τζέιμς έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ για, το, για την έκθεση, για το κείμενο. Φαίνεται ότι εξετάζουμε παλιά θέματα, όπως είπες George ε, ελπίζω να μην σε ενοχλεί που χρησιμοποιώ το μικρό όνομα. Δεν υπάρχει να βάση στις συνθήκες. Έχουν αποτύχει 60 πρωτοβουλίες και δεν δέχεται την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτές τις πρωτοβουλίες όταν παραβιάζει την περιοχή της, δεν της φύστης. Σου εύχομαι καλή τύχη με αυτά που περιέγραψες, παρόλο που δεν φαίνονται θετικά τα πράγματα. Έχω κάποια σοβαρή ανησυχία που την ετόπισες. Αφορά ε, την ψυχιακή ταυτότητα, την πανευρωπαϊκή Έχω πολύ σοβαρέ ανησυχίε περί αυτού, πιθανότατα διότι είχα εμπλακεί ε, σε κάποιες σε κάποια πολύ μεγάλα τέτοια προγράμματα ε, της ε, τεχνολογίας και τίθεται το πρόβλημα τη κυβερνοασφάλειας. Ίσως την έκθεσή σου μπορούσε να διασκεδάσει κάποιες ανησυχίες. Ε, με την πάρο του χρόνου να διασκεδάσει ανησυχίε που εκφράζω. Πού καταχωρούνται ε, τα άτομα και πού θα χρησιμοποιούνται αυτά τα στοιχεία. Θα είναι υποχρεωτική καταχώρηση για ταυτότητα για κάθε πολίτη ε, και θα υπάρχουν περιορισμοί όσον αφορά θέματα στα οποία θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτή ε, η ταυτότητα και σε τι θα μπορούν να ψηφίζουν. Θεωρείς ότι έτσι μπορεί να παρακαμφθούν διάφορα δημοψηφίσματα εθνικών κοινοβουλίων και αυτό είναι ο μεγαλύτερος φόβος μου ε, διότι επικεφαλής του Πρασίνου Κόμματος πέρσι προσπάθησε να απαγορεύσει πέρσι τα εθνικά δημοψηφίσματα. Αυτά τα σημεία, αν μπορείς να τα καλύψεις το έργο που επιτελείς, αυτό θα με βοηθούσε ούτως ώστε να μπορέσω να κατανοήσω ακριβώς τι προσπαθείς να επιτύχεις και κατά πόσο πραγματικά αυτό έχει κάποιο μέλλον, αυτή η όλη προσπάθεια κατά το τομέα. Συνάδελφος Χάρινγκ. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος κυρία Πρόεδρε. Να πω μόνο πως ε, Θεωρώ πως η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων θα πρέπει να προετοιμάσει το χρονοδιάγραμμα έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή του χρόνου να καταθέσει ένα νέο κανονισμό. Οπότε η πρωτοβουλία του συναδέλφου Τζόρτζ είναι πραγματικά απαραίτητη. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε η πρωτοβουλία αυτή η οποία τόσο συναισθηματικά φορτισμένη ήταν να καταλήξει σε πολιτική αποτυχία. Νομίζω ότι υπάρχει μια λύση και θα πρέπει να αναγνωρίσουμε πως αυτό το οποίο κάποτε παρουσιάσαμε ως μια νέα σχέση μεταξύ Ευρωπαίων πολιτών και Ευρωπαϊκής Ένωσης από την εμπειρία που έχουμε αποκτήσει τελικά απέτυχε. Οπότε είναι σημαντικό εμείς να παρουσιάσουμε μια πρόταση τροποποίησης του κανονισμού κατευθείαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να το κάνει του χρόνου πλην ε, λήξει η θητεία αυτή. Και για τα προηγούμενα θέματα τα οποία σχολιάστηκαν, ναι, συμφωνώ με όλα και με τις ε, αλλαγές προτείνει ο κύριος Σόφλεν και με τα όσα είπε η Σίλβια. Νομίζω όμως πως ε, για τον κανονισμό, για το σύστημα ε, ηλεκτρονικής ηθαγένειας Ευρωπαϊκής Ένωσης, νομίζω ότι θα πρέπει εδώ να εγκρίνουμε κάποιες από τις προτάσεις που κάναμε ε, στο κείμενο για την ηλεκτρονική δημοκρατία ή democracy. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε μια καλύτερη λειτουργία του συστήματος και γι' αυτό προτείνω στον Τζόρτζ κάποιες από τις ιδέες που είχαμε εκεί, που τις εγκρίναμε στην γνωμοδότηση για την ηλεκτρονική δημοκρατία, να τις εντάξει και στο δικό του κείμενο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Ράμον. Και πριν δώσω το λόγο στον Τζόρτζ, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι έχουμε προτείνει στα πλαίσια του προϋπολογισμού πιλωτικά προγράμματα. Ένα από αυτά είναι νέα τεχνολογία και εργαλεία πληροφορικής για την απλούστευση των πρωτοβουλειών των ε, πολιτών και πήραν πολύ ψηλό βαθμό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα αυτό το πρόγραμμα να υλοποιηθεί. Πριν δώσω το λόγο, είναι παρούσα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καμία φορά είναι εδώ. Όχι. Όχι. Τζόρτζ, ε, λοιπόν, έχεις ένα δίλεπτο για να ολοκληρώσεις το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ όλους τους ε, συναδέλφους. Χρησιμότατα και πολυτιμότατα τα σχόλιά σας. Και περιμένω τις τροπολογίες σας. Ψηφίζουμε 11 Οκτωβρίου. Και είναι πιο κοντά αυτή η ημερομηνία από ό,τι νομίζετε. Διότι θα απουσιάζουμε και περικατές εβδομάδες. Κάποιες σκέψεις δεν μπορώ να εξετάσω κάθε ενδεχόμενο. Για την ηλικία των 16 ετών είμαι ουδέτερος επ' αυτού. Επουδενή ε, δεν είμαι αντίθετος, αλλά γνωρίζω ότι υπάρχει μεγάλη αντίθεση όσον αφορά τη μείωση της ηλικία στο Συμβούλιο και θα πρέπει να δοθεί μάχη. Ε, είναι σημαντικό θέμα, αλλά δεν νομίζω ότι είναι και το σημαντικότερο. Αυτό, αυτά που είπε η κυρία Μπάρμπαρα Σπινέλη είναι πολύ σωστά, θα τα λάβω υπόψη. Για την Diane James έχω να πω κάποια πράγματα στην Diane. Τα ψηφιακά προβλήματα είναι σε μια φάση που δεν καταλαβαίνουμε ακόμα όλες τις συνέπειες, κυρίως τα θέματα ασφαλείας. Ήμουν στο Ταλίν. Μου είπαν ότι ο ψηφιακός κόσμος είναι υπέροχος. Δεν με τον θυσιασμό του σε τέτοιο βαθμό. Αυτή τελικά η ψηφιακή θα γίνει, δεν πρέπει να είναι υποχρεωτική, θα χρειαστεί χρόνος για να γίνει κάτι τέτοιο, θα πρέπει να είναι προαιρετική εφαρμογή και δεν θα πρέπει να παρακάμπτονται εθνικά δημοψηφίσματα ή ουδήποτε είδους δημοψηφίσματα. Όπως προσπαθώ να πω, αυτό δεν είναι άμεση δημοκρατία, είναι κάπου ανάμεσα ήμι άμεση δημοκρατία εμπλέκονται οι πολίτες σε σημαντικό ε, βαθμό, αλλά υπάρχουν πολλά σημεία δίθησης. Ευχαριστώ όλους ε, για την υποστήριξή τους, για τις προτάσεις τους και προσβλέπω στις τροπολογίες σας. Ευχαριστώ πολύ, George. Να σας πω τώρα ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα στον αυτό το θέμα. Προθεσμία υποβολή τροπολογιών, 5 το απόγευμα στις 8 Σεπτεμβρίου. Έχετε όλο το καλοκαίρι να το σκεφτείτε το θέμα. 8 Σεπτεμβρίου 5 το απόγευμα, συζήτηση 28 Σεπτεμβρίου και ψηφοφορία ελπίζουμε στις 11 Οκτωβρίου στην ε, Επιτροπή. Σας ευχαριστώ πολύ. Μπορούμε να πάμε στο σημείο 4 της διάταξης. Η σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όπως θα θυμόσαστε έχουμε δύο εισηγητές ε, για αυτό το θέμα. Για το ΕΛΚ έχουμε εμένα και για τους σοσιαλιστές τον Πέδρο Σίλβα Περέιρα Ίσως να μιλήσω εγώ για δύο λεπτά και να δώσω το λόγο μετά στον Πέντρο. Να σας πω ότι πρόκειται περί δυσχερέστα του ε, ζητήματος από πολλές πλευρές ε, για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά αυτή τη φορά έγινε ακόμα πιο δύσκολο το θέμα λόγω των προβλημάτων που δημιουργούνται από το Brexit. Και η ασφάλεια δικαίων το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ε, είναι ένα θέμα αυτό, οι εκλογές στο Ευρωκοινοβούλιο είναι ένα θέμα που απαιτεί απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αρκετά έγκαιρα, ώστε ε, τα διάφορα κράτη-μέλη με τι διάφορε νομοθεσίε να έχουν χρόνο να προετοιμάσουν όλε τι αναγκαίε νομικέ πράξει για τη διαδικασία και γι' αυτό επεξεργαστήκαμε το θέμα. Βέβαια, Καταλάβαμε από αυτά που είπε το Συμβούλιο ότι το αργότερο πριν το καλοκαίρι του χρόνου θα πρέπει να λάβει απόψη το Συμβούλιο. Θα πρέπει σαν Κοινοβούλιο να παρουσιάσουμε την έκθεση. Κανονικά πρέπει να την παρουσιάσουμε μέχρι το τέλος του προηγούμενου έτους. Αλλά για πάνω από ένα χρόνο αυτό το ζήτημα έχει παγώσει στη διάσκεψη των Προέδρων. Και αυτό παρά την αρχική μας ε, ε, δραστηριότητα και μετά την κοινοποίηση, ενεργοποίηση ε, του άρθρου 50 από την κυρία Μέη πάγωσε το θέμα και τώρα ε, γι' αυτό έχουμε περισσότερες χρονικές πιέσεις που ασκούνται πάνω μας να σας πω και κάτι άλλο όσον αφορά τη διαδικασία της προετοιμασίας του κανονισμού ότι Ήρθαμε σε επαφή με σχεδόν όλα τα κάτι μελη Ερχόταν εδώ μικρές και μεγάλες ομάδες εκπροσώπων ε, που ακολουθούσαν διαφορετικές προσεγγίσεις. Χρησιμοποίησαμε και τις απόψεις των εμπειρογνωμών. Θυμόσαστε τον Ιανουάριο. Έγινε μια μεγάλη ακρόαση με τη συμμετοχή μεγάλων εμπειρογνωμόνων που στα βιογραφικά τους έδειχναν ότι είχαν μεγάλη εμπειρία όσον αφορά την επεξεργασία των καταλήλων προσεγγίσεων που σχετίζονται με την απόφαση πρέπει να λάβουμε για τη σύνθεση του Κοινοβουλίου. Οπότε εδώ βρισκόμαστε σήμερα με όλες αυτές τις προκλήσεις, τα μισά του δρόμου. Πρόθεσή μας σήμερα είναι καταρχάς να ακούσουμε τις απόψεις σας. Πώς βλέπετε σήμερα μετά τις προηγηθήσεις συζητήσεις, πώς βλέπετε τα προβλήματα, ποια είναι τα σημαντικότερα για σας ζητήματα. Θα ξεκινήσω δίνοντας το λόγο στον Πέδρο και μετά θα δώσω και άλλες πληροφορίες για ζητήματα που θεωρώ σημαντικά που ίσως να μην καλυφθούν πλήρως από τον Πέδρο. Πέδρο, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, έγιναν αναλυτικές διαβουλεύσεις που πιστεύω ότι πρέπει να συνεχιστούν κάποιο διάστημα ακόμη για να επιτύχουμε ευρύτερη συνένεση για την πρότασή μας. Αλλά πώς έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Πολιτικά, βεβαίως, οι διαβουλεύσεις επιβεβαίωσαν αυτό που ξέραμε, ότι είναι πολύ λεπτό πολιτικά το θέμα. Κανείς δεν θέλει να χάσει έδραση. Και ιδιαίτερα τώρα που σε πολλά κράτη-μέλη γίνεται αντιληπτό ότι θα γίνει αναδιανομή κάποιων Βρετανικών εδρών. Άρα δεν μπορούμε να πείσουμε ότι πρέπει να μειωθούν οι έδρες. αλλά καμία ουσιώδης πρόοδος ε, προς την φθήνουσα αντιπροσπευτικότητα δεν είναι δυνατή σε αυτές τις συνθήκες. Και θα πρέπει να γίνει κάποια λοιπόν προσθήκη εδρών από τις έδρες του Ηνωμένου Βασιλείου. Επίσης ε, πρέπει να υπάρξει όσο ταχύτερα γίνεται νομική βεβαιότητα. Πρέπει λοιπόν να εγκριθεί η νομοθεσία έγκαιρα για να μπορέσει να εφαρμοστεί στις επόμενες ευρωεκλογές. Στα πλαίσια αυτά θεωρούμε ότι είναι δύσκολο να εγκριθεί μία μόνιμη ρύθμιση. Επιπλέον, σε πολλά κράτη-μέλη θεωρείται ότι υπάρχει σύνδεση μεταξύ της εκπροσώπησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το, το σύστημα ψηφοφορίας στο Συμβούλιο για να λήξει το σύστημα ψηφοφορίας στο Συμβούλιο πρέπει να γίνει αλλαγή των συνθήκων. Άρα μια μόνιμη ρύθμιση δύσκολο να επιτευχθεί. Όμως τελικά θεωρούμε ότι είναι δυνατόν να υπάρξει μια νέα ρύθμιση για την κατανομή των εδρών, μια μερική αναδιανομή των εδρών του Ηνωμένου Βασιλείου, μάλιστα θα έλεγα ενό ελάχιστου αριθμού εδρών του Ηνωμένου Βασιλείου, ούτως ώστε κανεί να μην χάσει έδρε. Και σε πλήρη συμμόρφωση με τις αρχές της συνθήκης της Λισαμβόνα. Δηλαδή πρέπει να βρούμε μία λύση που να εξασφαλίζει τη φθήνουσα αντιπροσωπευτικότητα, φθήνουσα αναλογικότητα. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξει ουσιώδης μείωση του αριθμού μελών του Κοινοβουλίου για να έχουμε περιθώριο απόδοση εδρών και σε περίπτωση μελλοντικών διευρύνσεων και για τις προτάσεις διεθνικών ψηφοδελτίων. Για τα θέματα αυτά χρειάζεται περαιτέρω συζήτηση. για να δούμε πόση στήριξη υπάρχει για αυτές ε, τις προτάσεις για διεθνικά ψηφοδέλτια, τι μορφή θα είχαν και ποιο θα ήταν το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ε, τέτοιων προτάσεων. Αυτά λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα. μπορούμε νομίζω να καταλήξουμε σε μια λύση που να βασίζεται σε αρχές που να συμμορφούνται πλήρως προς τις συνθήκες αλλά σε αυτή την περίπτωση θα χρειαστεί να διαθέσουμε κάποιες από τις έδρες του Ηνωμένου Βασιλείου. Τώρα, Υπάρχουν και τα προβλήματα του χρονοδιαγράμματος του Brexit. Και η λύση θεωρούμε ότι θα έπρεπε να είναι να διατηρηθεί το status quo κατανομής των θέσεων μέχρι, τη συμφωνία, μέχρι την έναρξη ισχύως της συμφωνίας αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου. Μόλις τεθεί σε ισχύ η αποχώρηση, τότε θα, θα υπάρξει αμέσως ένα νέο σύστημα κατανομής εδρών. Και αν η συμφωνία αποχώρησης συμβεί πριν από τις ευρωεκλογέ, δεν ξέρω τι θα γίνει, αλλά αν γίνει μετά θα έχουμε αυτομάτως το νέο σύστημα. Θα αρχίσει να ισχύει το νέο σύστημα. Α, αυτή είναι η κατάσταση χρειάζεται περαιτέρω συζήτηση για να υπάρξει ευρύτερη συμφωνία από αυτού και ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Υπάρχει ένα θέμα στο οποίο θα ήθελα να σταθώ. Είναι η σχέση αυτού του φακελού με ένα φάκελο που βρίσκεται εδώ και δύο χρόνια στο Συμβούλιο. Είναι ο εκλογικό νόμο και θα θυμόσαστε ίσω το άρθρο στη συνθήκη που αναφέρει πω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έπρεπε να προτείνει θα έπρεπε να καταθέσει μια πρόταση για τις ε, εκλογές, για την εκλογή προς το Ευρωκοινοβούλιο. Εμείς στην Ολομέλεια το εγκρίναμε το κείμενο αυτό το 2015 και το στείλαμε στο Συμβούλιο. Έκτοτε το δουλεύουν οι Προεδρίας και Νομίζω ότι στο σημείο αυτό θα πρέπει να σταθούμε γιατί αν πρόκειται να έχουμε αυτές τις ε, διασυνοριακές εκλογικές λίστες θα πρέπει να μπορούμε και εμείς να σας ενημερώσουμε ποιες θα είναι οι νομικές προϋποθέσεις που θα ισχύουν γιατί εάν θέλουμε στη σύνθεση του Ευρωπαϊκού ε, Κοινοβουλίου να έχουμε και τέτοιου είδους ε, ψηφοδέλτια θα πρέπει να το κάνουμε μέσω του εκλογικού νόμου που αποτελεί την μόνη νομική βάση που μας επιτρέπει κάτι τέτοιο. Το Συμβούλιο, δηλαδή τα κράτη-μέλη, στις συζητήσεις που κάνουν ε, επί της δικής μας πρότασης έχουν απορρίψει αρκετά σημεία. Το ένα ήταν το candidate, δηλαδή ο επικεφαλής ε, του ψηφοδελτίου και είπαν πως το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα δεν επιτρέπει κάτι τέτοιο. Νομίζω αυτό απηχεί το φόβο τους πως δεν θα μπορούσαν να επηρεάσουν αυτά τα ψηφοδέλτια και δεν θέλουν περισσότερη Ευρώπη στο σημείο αυτό. Και η πρόκληση που αντιμετωπίζουμε σήμερα είναι το κατά πόσο μπορούμε να προχωρήσουμε και στο θέμα της σύνθεσης του Κοινοβουλίου, αλλά και το κατά πόσο υπάρχει αυτή η πλειοψηφία για την ε, Ευρωπαϊκή Εκλογική Περιφέρεια και κατά πόσο αυτό μπορεί να μας βοηθήσει στο να πείσουμε ε, το Συμβούλιο να κάνει κάτι παραπάνω για τον εκλογικό νόμο. Θα τα δούμε αυτά και νομίζω ότι πρέπει να γνωρίζετε ακριβώς ποια είναι τα θέματα που συζητιώνται. Επίσης, ο τρόπος με τον οποίο θα λειτουργεί αυτός, αυτό το ψηφοδέλτιο και το κατά πόσο η εκλογή αυτή θα γίνεται παράλληλα ταυτόχρονα με τις εθνικές εκλογές για τα εθνικά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οπότε και τα θέματα αυτά πρέπει να λυθούν. αυξάνοντας τον κατάλογο των δυσκολιών που θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε με το φάκελο. Έχουμε μπροστά μας μισή ώρα. Θα ήθελα να μου πείτε ποιοι θέλετε να μιλήσετε. Ξέρω πως είναι οι σκιώδες. Αφήνω και τους υπόλοιπους. Ο Παύλο Καστάλτο δεν είναι εδώ, αλλά δεν υπάρχει αντικαταστάσεις. Αντικαταστάτης. Κύριο κύριος δεν ξέρω αν κάποιο άλλος θέλει να προσθεθεί στον κατάλογο ομιλητών. Πρέπει να κλείσω τον κατάλογο ομιλητών για να αποφασίσω μετά πόσο χρόνο θα σας διαθέσω. Δεκατρεις θέλουν να λάβουν το λόγο, υπάρχει άλλος. Κλείνει ο κατάλογος, λυπούμε γι' αυτό. Δεκατρεις ομιλητές. Σχεδόν δύο λεπτά ο καθένας. Εστέλα Κονική λοιπόν, παρακαλώ. Και σαφής. Κυρίως για το θέμα των ε, περιεθνικών αυτοκαταλόγων καταλόγων και οτιδήποτε άλλο θέλετε να θίξετε. Αλλά θέλουμε να δούμε ποια είναι η άποψή σας ε, για την κατανομή των 73, το πιο δύσκολο θέμα πρέπει να έχουμε μια ομαλή προσγείωση για τα κάτι μελη που θα χρησιμοποιήσουν αυτή τη λύση ε, και όσον αφορά την ε, φθήνους αναλογικότητα. Λοιπόν, αυτά τα ζητήματα. Αυτά τα ζητήματα λοιπόν. Κλείνει ο κατάλογος. Δύο λεπτά ο καθένας παρακαλώ. Κανένας μετά τον Ραμόν Χαουρέγγι. Ο κ. Βιασδόφσκι είναι ο πρώτος που έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα είμαι πολύ σύντομος. Πάντα εγώ είχα δισταγμού όσον αφορά την κατανομή των εδρών, διότι το Ηνωμένο Βασίλειο εξακολουθεί να παραμένει μέλος και ίσως ε, να είναι ακόμα μέλος και την Άνοιξη και το καλοκαίρι του 2019. Όμως, Εάν πρόκειται να γίνει διανομή, κατανομή των εδρών, η πιο λογική θέση θα ήταν ο μηχανισμός του Cambridge, στη βασική μορφή που έχει. Αυτό είναι κάτι που συστήνω. Το Συμβούλιο δεν είναι ικανοποιημένο όσον αφορά αυτούς τους υπερεθνικούς καταλόγους. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε την εφαρμογή του παλιού συστήματος, όσον αφορά την όλη ιδέα εγώ θα συνέστηνα το συμβιβασμό του Cambridge. Προφανώς περιμένω τις συζητήσεις και πιστεύω ότι όλοι περιμένουν για κάποιες προτάσεις και συστάσεις από πλευράς των εισηγετών. Ευχαριστώ κύριε Φερχόφστατ. Πολύ σύντομα, ευχαριστώ πολύ τους δύο συγητές. Είναι σοφή αυτή η συμβουλή που μας δίδεται να συνδυάσουμε και τα δύο θέματα, δύο με το Συμβούλιο αργότερα, θα έχουμε συνδυασμό ε, συνθέσεως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εκλογικών νόμο, από την άλλη. Είναι οι δύο ε, όψεις του ιδίου προβλήματος θα έλεγα. Αν επιτρέπετε, Πρόεδρε, εγώ θα έλεγα το εξής. Στην έκθεση να αναφέρουμε τρεις αρχές η πρώτη. Εάν συμβεί το Brexit, έχουμε καταρχήν την, ε, τη βασική αρχή της μειώσεως των εδρών. Όλοι θα κατανοούν ότι είναι κάτι αναγκαίο. Όταν μια μεγάλη αντιπροσωπεία ε, ε, με 73 έδρες αποχωρεί από το Κοινοβούλιο. Μετά είναι αυτή η φθήνουσα αναλογικότητα. Εκεί να μην πούμε ότι κανένα κάτω μέλος δεν μπορεί να χάσει έδρα. Ε, δεν έχει συμφέρον το κοινοβούλιο αυτό να το συμπεριλάβει ρητά στην έκθεση. Ίσως εκεί να καταλήξουμε. Και είναι ρεαλιστικό αυτό να καταλήξουμε εκεί αν έχουμε κάποιο είδους ε, φθήνουσα αναλογικότητα. Μη το συνδέσουμε με στο θέμα με τη φθήνουσα λογικότητα. Διότι αν δεν συμπεριληφθεί αυτό ενισχύει τη θέση του Κοινοβουλίου. Θα πρέπει αυτό να το αξιώσουν τα κράτη-μέλη. Να μην είναι όμως μια βασική αρχή που θεσπίζουμε την αρχή. Και άλλη αρχή, η τρίτη. Αυτό με, τους με τα ευρωπαϊκά ψηφοδέλτια, η ευρωπαϊκή δημοκρατία θα έπρεπε να είναι δυνατό. Αυτό που δεν ήταν δυνατό στον εκλογικό νόμο του 2015, διότι δεν είχαμε το Brexit, γίνεται εφικτό μετά το Brexit. Δηλαδή, να βρούμε μια ισορροπία μεταξύ μειώσεως των εδρών, φθήνουσας αναλογικότητας και των ε, ευρωπαϊκών αυτών ε, ψηφοδελτίων. Εγώ τι θα έλεγα, Πρόεδρε, να μην προχωρήσουμε πολύ γρήγορα διότι πράγματι αληθεύει ότι χρειάζονται κάποιο χρόνο να προσαρμόσουν τις νομοθεσίες τους ε, τα κάτι μελη Αλλά αυτό είναι και ένα εργαλείο και για μας. Και είναι πολύ σημαντικό να το λάβουμε υπόψη αυτό το στοιχείο. Απαιτείται συμφωνία με το Συμβούλιο. Θα είδατε ότι σε κάποια κράτη-μέλη υπάρχει μια συγκεκριμένη στάση όσον αφορά την ευρωπαϊκή δημοκρατία και τα ευρωπαϊκά ψηφοδέλτια. Αλλάζει η στάση δραματικά και γρήγορα και προσθετική κατεύθυνση. Τέλος, να υπογραμμίσω κάτι. Το θέμα της Ιρλανδίας και της Βορείου Ιρλανδίας. Στο μέλλον θα υπάρξουν 500.000, 600.000 Βόρειο Ιρλανδοί με Ιρλανδικό διαβατήριο. Αυτοί οι άνθρωποι θα είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα, κατά την άποψή μου, να συμμετέχουν στις ευρωεκλογέ. Ακόμα και όταν δεν ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά στη Βόρεια Ιρλανδία. Αλλά κατέχουν Ιρλανδικό ε, διαβατήριο και Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια. Η αδίποτε κατανομή των εδρών πρέπει να λαμβάνει υπόψη αυτό το πρόβλημα με συμπληρωματικέ έδρε για την ε, Δημοκρατία τη Ιρλανδία, κατά την απόψη μου. Ε, πράγματι, η Δημοκρατία τη Ιρλανδία είναι κατά τη ιδέα να δώσει τα δικαιώματα αυτά στου υπηκόου τρίτων ε, χωρών να ψηφίζουν. Οπότε έχουμε ένα πρόβλημα. Και κάτι άλλο να πω. Μιλήσατε αναφερθήκατε στο παιχνίδι του χρόνου. Παίξαμε το χρόνο επί μακρόν, διότι η απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την πρόταση του Ευρωκοινοβουλίου έδωσε μια προθεσμία που παρήλθε το περσινό Δεκέμβριο. Οπότε ήδη παίζουμε με το χρόνο. Ευχαριστώ για τη συμβουλή σας. Μπορούμε να προχωρήσουμε. Στον κύριο Σόλτς. ότι έχεις το λόγο. Δύο λεπτά παρακαλώ, ώστε να καλύψεις και αυτά που, το χρόνο που πήρε παραπάνω εκεί. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο σύντομο γίνεται. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας πρέπει να αντιμετωπίσουμε το περίπλοκο χαρακτήρα των προβλημάτων. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι η κατανομή των εδρών κατά κάποιο τρόπο σχετίζεται με τον λογικό νόμο. Συζητούμε ότι έχει μπλοκαριστεί το θέμα του εκλογικού νόμου στο Συμβούλιο. Σημειώνουμε αυτά που μας είπατε για τη θέση του Συμβουλίου. Αργότερα μπορούμε να το συζητήσουμε εδώ πρέπει να είμαστε πολύ πιο θαραλέοι, ειλικρινείς και διαφανείς σχετικά με τις επιθυμίες μας για τον εκλογικό νόμο. Όσον αφορά την κατανομή των εδρών, πιστεύω ότι θα πρέπει το τέλος του έτους να έχουμε κάποια θέση. Τα κράτη-μέλη να μπορούν να προωθήσουν τη λύση στην εθνική τους νομοθεσία. Θα πρέπει να ετοιμαστούν για τις εκλογές. Γι' αυτό εγώ θα προειδοποιούσα. Θα έλεγα ότι κατανέμουμε ήδη τις έδρες του Ηνωμένου Βασιλείου και ρυθμίζουμε κάποια θέματα και αυτό μπορεί να είναι αρνητικό μήνυμα για τις διαπραγματεύσεις. Κανείς δεν ξέρει ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων του Brexit και γι' αυτό θα έλεγα ναι θα πρέπει να συμπεριλάβουμε την αρχή της κατανομής των εδρών αν λάβει χώρα το Brexit αυτό πρέπει να είναι κατανοητό της πάση και θα πρέπει Επίσης, να αποφασίσουμε για τη μέθοδο. Εγώ είμαι υπέρ των ευρωπαϊκών ψηφοδελτίων. Ε, η ομάδα μου έχει διαφορετικές απόψεις επ' αυτού, αλλά πρέπει να το συζητήσουμε περαιτέρω, διότι νομίζω ότι στην κατάσταση που βρισκόμαστε θα πρέπει να δούμε ποιο τρόπο μπορούμε να ενισχύσουμε περισσότερο την ιδέα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως πώς θέλουμε να έχουμε τη νέα ευρωπαϊκή προσέγγιση και αντίληψη, να δώσουμε περισσότερο λόγο στους πολίτες. Τέλος, στηρίζω το έγγραφο εργασίας σας. Να χρησιμοποιήσουμε τις διακοπές της θερινές για να απαντήσουμε στα τρία ερωτήματα στο τέλος του εγγράφου. Μας δίνεται τη δυνατότητα να επεξεργαστούμε κάποιες πτυχέ και ίσως στις συζητήσεις του Σεπτεμβρίου θα πρέπει να καταλήξουμε σε κάποια θέση. Πασκάλ Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πολύ σύντομα γιατί έχουμε χρονική πίεση. Να απαντήσω και στον Γκί Φερχόφστατ. Υπάρχει πραγματικότητα, έχουμε διάφορες δυνατότητες και να δούμε τι πραγματικά θα συμβεί. Τι θα πραγματικά συμβεί. Βεβαίως θέτουμε την αρχή της φθήνουσας αναλογικότητας Βεβαίω πρέπει να το κάνουμε και ξέρουμε ότι αν δεν αξιοποιήσουμε τις 73 βρετανικέ έδρε, έδρες, κάποια κράτη-μέλη θα έχαναν έδρε. Άρα φυσικά θα τον μπλοκάρουν στο Συμβούλιο. Άρα για μια φορά θα είμαι πιο πραγματιστή από τον Γκί. Προτείνω, είναι μια πρόταση, προτείνω να αξιοποιήσουμε το γεγονός ότι θα φύγουν οι 73 έδρες για να εφαρμόσουμε επιτέλους και οριστικά την αρχή του Cambridge. Θα επέτρεπε λοιπόν οι μέσου ε, μεγέθους χώρες να έχουν περισσότερες έδρες και να μιλήσω και ως Γάλλος, κάτι που δεν κάνω ως Ευρωβουλευτής, στη Γαλλία ε, ως φεντεραλιστής θεωρώ ότι έχουμε την τύχη να έχουμε έναν πρόεδρο φεντεραλιστή που έχει θέσει το θέμα των διεθνικών ψηφοδελτίων στο πρόγραμμά του. Ποτέ δεν είχε γίνει αυτό στη Γαλλία. Είναι μια πρόοδος αυτό. Και θα ήθελα, εφόσον ο συμβασμός του Κέμπριους μας επιτρέπει να ε, διαθέσουμε 28 έδρες, μία αναχώρα. Δεν είναι αυτό που ζητώ για, τις διεθνικές, για τα διεθνικά ψηφοδελτία. Να αξιοποιήσουμε αυτές τις 28 έδρες για να προωθήσουμε την αρχή των διεθνικών ψηφοδελτίων, να αξιοποιήσουμε το βάρος της Γαλλίας στο Συμβούλιο για να υπάρξει πρόοδος του θέματο αυτού. Αυτά εντάχει. Ευχαριστώ. Γερόλφ Άνεμανς. Αγαπητοί συνάδελφοι, είχα ήδη πει ότι Βεβαίως θα πρέπει να μειωθεί ο αριθμός των εδρών, αλλά πρέπει όλοι να συμφωνήσουν. Το Brexit πρέπει να έχει την επίπτωσή του και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Διότι νομίζω ότι έχει υπάρξει περισσότερος ενθουσιασμός μετά το Brexit για την φεντεραλιστική προσέγγιση. Πρέπει λοιπόν να αρκεστούμε σε λιγότερες έδρες ο συνάδελφος Φερχόφστατ. Βεβαίως ξέρω ότι είναι ιδιαίτερα υπέρμαχος των διεθνικών σφοδελτίων. Νομίζω όμως, όμως εμείς δεν είμαστε τόσο ενθουσιώδεις. Θα πρέπει νομίζω να περιοριστούμε σε λιγότερες έδρες συνολικά. Ευχαριστώ πολύ. Ο Γιώ Λάινεν. πιστεύω ότι πρέπει να βασιστούμε στην πολιτική πραγματικότητα. Το άρθρο 50 έχει ενεργοποιηθεί που προβλέπει δύο χρόνια για την αποχώρηση μιας χώρας. Άρα η Βρετανία το Μάρτιο του 19 με βάση ό,τι γνωρίζουμε θα πρέπει να αποχωρήσει. Άρα δεν θα συμμετάσχει στις επόμενες ευρωεκλογές. Αυτό διευκολύνει την εφαρμογή της φθήνουσας αναλογικότητας μέσω κάποιας διανομής των εδρών. Αλλά εγώ θα έλεγα ότι πρέπει να διανύμουμε ένα περιορισμένο αριθμό εδρών. Γιατί πρέπει να δράσουμε με υπευθυνότητα. Να δείξουμε ότι όσο μικραίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, μικραίνει και το Κοινοβούλιο. Δεν θα ήθελα να έχουμε πάνω από 700 έδρε. Η αναδιανομή λοιπόν να μην ε, υπερβεί και καλύτερα να είναι κάτω από τις 700 έδρες. Αυτό είναι και το μήνυμα ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ακριβώς προσαρμόζεται στη νέα ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Τώρα βέβαια έχουμε 751 έδρες. Άρα θα πρέπει να αναφέρουμε και τα διεθνικά ψηφοδέλτια. Είναι αυτό κάτι που το Κοινοβούλιο το λέει εδώ και 20 χρόνια. Υπενθυμίζω ότι η συνθήκη της Λισαβόνας λέει ότι εκπροσωπούμε τους πολίτες της Ένωσης. Όχι απλώς τους πολίτες ε, του κράτους μέλους μας. Κατά τη γνώμη μου λοιπόν και ο εκλογικός νόμος και η σύνθεση του Κοινοβουλίου δεν εκπροσωπούν τη συνθήκη της Λισαβόνας πλέον. Συμφωνήθηκαν τον προηγούμενο αιώνα. Πρέπει να έχουμε λοιπόν και εθνικά ψηφοδέλτια και διεθνικά ψηφοδέλτια. Αλλά Υπάρχει ένα déjà vu από τον εκλογικό νόμο. Το Συμβούλιο πρέπει να αποφασίσει ομόφωνα και δεν αποφασίζει ομόφωνα. Αλλά αντίθετα από τον Σνάλφο Γιζαντόφσκι που λέει ότι δεν θα χάρει το Συμβούλιο, δεν νομίζω αγαπητέ Σνάλφε, ότι το καθήκον μας είναι να ευχαριστούμε το Συμβούλιο. Το ζήτημα είναι να είναι καλό το σύστημα. Να το αναφέρουμε αυτό. Λοιπόν, να καταλήξουμε μια θέση, θα διαπραγματευτούμε το Συμβούλιο και θα δούμε πού θα καταλήξουμε. Πρόεδρο. Μα δεν υπάρχει διαπραγμάτευση με το Συμβούλιο. Θα πρέπει στόχος μας να είναι να αποφασίσουμε κάτι το οποίο να μπορεί να εγκρίνει το Συμβούλιο. Ναι, λέει ο κύριο Λάινεν, αλλά πρέπει να το αποδεχθούμε και εμεί στο τέλο. Έλμαρ Μπροκ. Νομίζω ότι η διατύπωση του Τζο Λάινεν ότι το σύστημα πρέπει να είναι καλό, ε, είναι σοσιαλιστική διατύπωση. Μάλιστα τα, οι λέξεις που χρησιμοποίησε είναι ότι πρέπει να είναι χαρούμενο το σύστημα, μόνο οι σοσιαλιστές μπορούν να είναι τέτοια πράγματα. Τώρα σοβαρά τώρα. Ε, ανέφερε στο θέμα με τον ε, επικεφαλής ψηφοδελτίων. Α, δεν είναι υπόρρο συζήτηση, αλλά θα πρέπει να το συζητήσουμε. Θα πρέπει να... ε, ε δεν θα πρέπει να ε, ε, το βάλουμε στο κείμενο γιατί αυτό θα σημαίνει περιορισμό. Το λέει η συνθήκη της Λισαβόνας πώς ε, καταρτίζουν τα ψηφοδέλτια. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να το συζητήσουμε με το Συμβούλιο. Έχουμε λοιπόν μια, μια θέση την οποία θα πρέπει να διευρύνουμε γιατί αν υπάρξουν νομοθετικέ ρυθμίσει θα αποδυναμωθεί η θέση μα. Και με βάση αυτά που συνέβησαν την προηγούμενη φορά στι εκλογέ, προεδοποιώ να μην το κάνουμε. Θα δώσουμε δυνατότητα στο Συμβούλιο να αρχίσει να κάνει ζημιά εκεί πέρα μέσα. Ξέρετε πολύ καλά πώ καθορίζει τον πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Συμβούλιο μετά από τη διαβούλευση με το Κοινοβούλιο και, ενώ, λαμβάνοντα υπόψη το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Λοιπόν, ή, ε, ε, δεν ξέρω αν είμαι ο που δεν είμαι τόσο πεισμένο για τα διεθνικά ψηφοδέλτια. Έχω δύο λόγου. Ξεκολουθώ να έχω δύο λόγου. Έχω την ε, παλιωμοδίτικη γνώμη ότι πρέπει να είμαστε κοντά στους ψηφοφόρους μας. Γιατί τον περισσότερο χρόνο είμαστε πολύ μακριά από τους ε, βουλευτές. Ας δούμε το βρετανικό και το ιρλανδικό σύστημα. Είναι καλύτερα από αυτά που έχουμε. Ο πολίτης πρέπει να καταλαβαίνει να αυτός είναι ο ευρωβουλευτής μου. Αν δεν γίνει αντιληπτό αυτό από τους πολίτες, έχουμε πρόβλημα της εγκύτητάς μας προς τους πολίτες. Άρα έχουμε θέμα νομιμοποίησης. Ως ε, Ευρωπαίο ε, Φεντεραλιστή καταλαβαίνω τα διεθνικά ψηφοδέλτια. Αλλά δεν μπορώ να το συνδέσω αυτό, να το συνδυάσω με το πρώτο σημείο. Αλλά ποιο κάνει την επιλογή τελικά για αυτά τα ευρωπαϊκά ψηφοδέλτια. Τα πολιτικά κόμματα. Πώς θα γίνεται. Πώς επιλέγονται. Και με ποια διαδικασία. Με ποια δημοκρατική διαδικασία θα το κάνει κάποιο σόφρον προεδρείο, θα υπάρχει ένα σύστημα συμμετοχής της βάσης. Στη Γερμανία, για παράδειγμα, μπορεί κανείς να γίνει ευρωβουλευτής μόνο αν επιλογεί μέσω μιας διαδικασίας, ε, μέσω του κόμματος. Όλα τα άλλα ε, είναι παράνομα. Όπως γίνεται σε άλλες χώρες, για παράδειγμα, που επιλέγεται από το Προεδρείο, για παράδειγμα, ενός κόμματος ή από τον αρχηγό. Υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία που προβλέπεται στη Γερμανία. Πρέπει να βρούμε απάντηση λοιπόν στο θέμα αυτό. Το δεύτερο. Έχουμε την κατανομή με βάση τα, τα κράτη-μέλη. Πώς θα υπάρχει κατανομή στα κράτη-μέλη σε διεθνικά ψηφοδέλτια. ίσως ε, να ευνοούνται οι υποψήφοι από τα μεγάλα κράτη, γιατί πολλοί θα ψηφίζουν, ε, θα σταυρώνουν τους ε, υποψήφιους από το κράτος μέλος τους. Άρα θα ευνοούνται οι υποψήφοι από τα μεγαλύτερα κράτη-μέλη. Αυτά είναι και τεχνικά θέματα, αλλά και πολιτικά θέματα. Όλα αυτά πρέπει να τα δούμε πριν αρχίσουμε να διατυπώνουμε τις επιθυμίες μας. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε 7 ομιλητές και 7 λεπτά. Ένα λεπτό ο καθένας και μετά θα σας κόβω. Θα πρέπει να αναλάβετε την ευθύνη για τους συναδέλφους σας. Πάουλο, Ράντζελ. Θα είμαι πολύ σύντομος. Είναι μια μεγάλων ε, διαστάσεων ευκαιρία να διορθώσουμε ορισμένα λάθη του παρελθόντος για να υλοποιήσουμε επιτέλους την αρχή της φθήνουσας αναλογικότητας. Πρέπει λοιπόν να το κάνουμε. Αλλά θα πρέπει να υπάρχει μια ρήτρα που να λέει και αυτή είναι νομίζω και η γνώμη των συνεισηγητών που να λέει λοιπόν ότι Εάν για οδήποτε λόγο ε, παραμείνει το Ηνωμένο Βασίλειο ή παραμείνει περισσότερο από ό,τι προβλέπεται, τότε η ρύθμιση αυτή θα αρχίσει να ισχύει όταν υπάρξει αποχώρηση. Αλλά νομίζω ότι νομικά αυτό γίνεται. Η μόνη μου ανησυχία ότι δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι τα 28 κράτη-μέλη θα εγκρίνουν την εκλογική νομοθεσία. Και αν δεν τους αρέσει η τελική λύση, μπορεί να μπλοκάρουν αυτή την ερήτρα Πρέπει λοιπόν και αυτό να το έχουμε υπόψη μας. Επίσης, για τα διεθνικά ψηφοδέλτια. Έχω συζητήσει με ευρωβουλευτές από μεσαίων διαστάσεων χώρες και ναι μένουν υπέρ της αρχής, αλλά δεν νομίζουμε ότι είναι τώρα η κατάλληλη συγκυρία γιατί είναι ήδη περίπλοκη διαπραγμάτευση και γιατί υπάρχει ο κίνδυνος ε, που ανέφερε ο Έλμαρ Μπρόκ. Είμαι πεπισμένος, γιατί ξέρω πώς λειτουργούν αυτά τα ζητήματα, ότι, ότι θα υπάρχει τελικά ενίσχυση των μεγαλύτερων χωρών. Για τις μικρομεσαίες χώρες αυτό δεν θα ήταν καλό. Δεν θα ήταν λοιπόν ευρωπαϊκά ψηφοδέλτια, θα ήταν τελικά εύνοια προς τις μεγαλύτερες χώρες. Γι' αυτό το λόγο δεν συμφωνώ. Μπορούμε το φέρουμε. Ευχαριστώ. Η κυρία Τζέιμς. Σύντομα παρακαλώ. Λοιπόν, να αναφερθώ σε δύο παρατηρήσεις του κυρίου Φερέιρα. Είπατε κάποιες έδρες του Ηνωμένου Βασιλείου. Και το δεύτερο σχόλιο σα όταν η συμφωνία σε τεθεί ενισχύ. Αυτές οι δύο προτάσεις λένε ότι εσείς φαίνεται ότι θεωρείτε ότι θα υπάρξει μια μεταβατική φάση μετά τον Μάρτιο του 19. Αν το επιβεβαιώσετε, θα μας βοηθούσε να καταλάβουμε μια άλλη απόχρωση που θα αναφερθεί για το θέμα αυτό. Αν το Ηνωμένο Βασίλειο είναι σε μεταβατική φάση, πότε θα είναι η καταληκτική ημερομηνία. Γιατί πρέπει να το δούμε και αυτό. Για το πώς θα συμμετέχουν οι συνάδελφοι. Και μία ρεαλιστική συζήτηση για το πώς θα συμβάλλουν. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει εγώ νομίζω ότι πρέπει να είμαστε είτε εντό είτε εκτός. Τώρα φαίνεται ότι ε, κάποιοι θέλουν να υπάρξει μεταβατική περίοδο και δεν βοηθάει αυτό. Ευχαριστώ η κυρία Τεπαρντέλ. Ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ σημαντικό θέμα για όλα τα κράτη-μέλη για τον Brexit. Πριν συζητήσουμε την κατανομή των εδρών, Πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι το 2019 θα έχει αποχωρήσει το Ηνωμένο Βασίλειο. Για να μπορέσουμε να πούμε θα διαθέσουμε τις έδρες τους. Δεν ξέρω θα γίνει κάτι τέτοιο. Αν όμως ε, ισχύει, τότε βέβαια μπορούμε να αναδιανύμουμε κάποιες έδρες. Αλλά έχουμε τις δύο αρχές, της φθήνουσας αναλογικότητας, αλλά παράλληλα είναι πολύ σημαντικό να προσθέσουμε και την δημογραφική αρχή, δηλαδή τον πληθυσμό της κάθε χώρας. Και σας το λέω χωρίς καμία αμφιβολία. Κανένα κράτος μέλος δεν θα θελήσει να αποδεχθεί μείωση των εδρών του. Κανένα κράτος μέλος. Δεν θα δεχθεί με βάση την αρχή της αναδιανομής να έχει λιγότερες έδρες από κάποιο άλλο κράτος μέλος που έχει λιγότερους κατοίκους. Πρέπει λοιπόν να βασιστούμε σε αυτές τις δύο αρχές. Τώρα για τα διεθνικά ψηφοδέλτια. Βεβαίως θα μπορούσε να εδραιώσει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά εάν δεν έχουμε σαφείς αρχές για το πώς θα καταρτίζονται αυτά τα ψηφοδέλτια και ποιους θα εκπροσωπούν, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε γιατί πρέπει η αρχή μας να είναι η ισότητα όλων των πολιτών και η δίκαιη εκπροσώπηση όλων των πολιτών. Περβάνος Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Με ενοχλούν τα δύο λεπτά που μου δώσατε γιατί αυτή η συζήτηση είναι θεμελιώδου σημασία. Το συζητάμε το θέμα αυτό εδώ και πολύ καιρό και είναι η πρώτη φορά που το συζητάμε. Ε, με κάπως συγκεκριμένη βάση. Οπότε σας παρακαλώ να μην με διακόψετε. Θα επιδιώξω να μην ε, μακρηγορήσω ιδιαίτερα. Γιατί έχω πολλά να πω. Πρώτον, για τον Brexit. Το Κοινοβούλιο σε όλα τα ψηφίσματα αναφέρει ότι είναι αποφασισμένο να συνεχίσει να ασχολείται με τις υποθέσεις που το αφορούν και να προωθεί την ε, ευρωπαϊκή οικοδόμηση σε όποια φάση και αν είναι η διαπραγματεύση για τον Brexit. Και συμφωνώ με τον συνάδελφο Γιολάνε. Το άρθρο 50 έχει ενεργοποιηθεί και μέχρι στιγμής το Brexit θα γίνει πριν τις επόμενες ευρωεκλογέ για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι καιρό λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, να ασχοληθεί με το θέμα αυτό για δύο λόγους. Γιατί το θέμα αυτό είναι θέμα εντός της εντολής του και το χρονοδιάγραμμα του Brexit μας υποχρεώνει. Δεύτερον, για το θέμα της φθήνουσας αναλογικότητας. Ευχαριστώ τους δύο συνεισηγητές που υπενθύμησαν την αρχή και που την έθεσαν ως βασική αρχή της έκθεσής τους. Είναι πολύ σημαντικό. Αν θέλουμε να υπάρξει μία βιώσιμη λύση. Πρέπει να αποφύγουμε να χάσουν τα κράτη-μέλη έδρες αν θέλουμε να υπάρχει κάποια πιθανότητα ομοφωνία στο Συμβούλιο. Αλλά δεν μπορούμε να εισάγουμε τώρα μια νέα αρχή. Την αρχή της ε, υπερφθήνουσας, της υπερβολικά φθήνουσας αναλογικότητας. Ελπίζω να καταλάβαν να εισαγουμε τωρα μια νεα αρχη την αρχη της υπερφθηνουσας της υπερβολικα φθηνουσας αναλογικοτητας ελπιζω να καταλάβανε ολοι τι εννοώ. Τρίτο θέμα. Βλέπω διάφορα νούμερα να κυκλοφορούν, τα οποία εφαρμόζουν αυτή την αρχή της υπερβολικής, υπερβολικά φθήνουσας αναλογικότητας. Κάτι άλλο που βεβαίως ε, συμφωνεί με τις ιδέες σας, αλλά δεν το αναφέρατε. Όλες οι προβλέψεις πρέπει να γίνουν με βάση τις πιο προ... Προ... απογραφές. Να έχουμε στοιχεία δηλαδή του 16. Επίσης είναι επίγον να προχωρήσει η Επιτροπή μας για το θέμα αυτό. Γιατί ξέρουμε ότι η απόφαση πρέπει να ληφθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Και έχει αρχίσει μια πολύ πιεστική αντίστροφη μέτρηση. Δεν ξέρω μήπως ε, ε, ε, θέλετε να αναβάλλετε ξέρω εγώ, τις ευρωεκλογές αλλά μέχρι στιγμής δεν το έχω ακούσει ίσως να γίνει και αυτό αλλά μέχρι στιγμής το θέμα του πότε θα υποβληθεί η έκθεση, πότε θα υποβληθούν τροπολογίες, πότε θα πάει στην Ολομέλεια. Δεν τα είπατε. Μα είναι θεμελιώδες αυτό. Νομίζω ότι αρχικά το, χρονοδιάγραμμα προέβλεπε ότι έπρεπε να ψηφίσουμε το Σεπτέμβριο. Νομίζω ότι ήδη έχει ξεπεραστεί αυτό. Επίσης, θα προτιμούσα να υιοθετήσουμε μια μόνιμη λύση. Είπατε όμως ότι υπάρχει πρόβλημα στο Συμβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να υιοθετήσει ω κοινοβούλιο, ω θεσμό την άποψή του. Δεν είναι τώρα δικό μα θέμα να προκαταλάβουμε ή να ε, ανησυχούμε για τους συναισθηματισμούς του Συμβουλίου και για τους εκνευρισμούς του. Πρέπει να ασκήσουμε τα καθήκοντά μας. Πρέπει να παρουσιάσουμε την άποψή μας για την κατανομή των εδρών και κατόπιν το Συμβούλιο θα υιοθετήσει τη δική του άποψη. Δεν ε, πρέπει εμείς ε, να ανησυχούμε για τις ανησυχίες του Συμβουλίου για τα διεθνικά ψηφοδέλτια. Βεβαίως ε, είμαι φίλη και θαυμάστρια του Άντζου Νταφ παρά τότε έχει αποχωρήσει από το Κοινοβούλιο και το θαύμαζε όσο ήταν συνάδελφο. <coughs> Είμαι υπέρ των διεθνικών ψηφοδελτίων. Και νομίζω ότι ε, υπάρχει κάποια στήριξη και από τα κράτη-μέλη. Αλλά δεν θα ήθελα να παγιδεύσει τη δυνατότητά μας να επιτύχουμε αυτό που είναι εφικτό, ιδιαίτερα για θέματα δημοκρατικότητας, γιατί το σημερινό σύστημα δεν είναι δίκαιο, άρα δεν είναι δημοκρατικό. Αλλά θέλω να θέσω το ερώτημα στους συνεισηγητές. Δεν θα υπήρχε δυνατότητα να υπάρξουν δύο προτάσεις. Μία για τη σύνθεση του Κοινοβουλίου και με την ελάχιστη δυνατή χρήση των Βρετανικών εδρών και επίσης μια άλλη πρόταση όπου το Κοινοβούλιο δεν, θα τα, συνδέ, δεν τα απόλυτα τα δύο γιατί αν τα συνδέσουμε τότε δίνουμε όπλα στο Συμβούλιο κάνουμε πολύ εύκολο κάποιος να σκίσει βέτο αυτή θα ήταν μια δυνατότητα να προχωρήσουμε ευχαριστώ που δεν με διακόψατε Ευχαριστώ πολύ. Ο Μάπς Άντερσον είναι ο επόμενος. Πιστεύω πως θα πρέπει να φανούμε πάρα πολύ προσεκτικοί και δεν θα πρέπει να θεωρήσουμε εκ των προτέρων πως θα έχει λάβει χώρα το Brexit πριν από τις επόμενες εκλογές. Μπορεί να σημειωθούν καθυστερήσεις. και δεδομένη της έλλειψης δεξιοτήτων τη κυβέρνηση των συντηρητικών μπορεί να μην γίνει τελικά το Brexit. Αυτό δεν είναι πολύ πιθανό, αλλά α μην κάνουμε υποθέσεις. Και αν καθυστερήσει, αν αποτραπεί, δεν θα έπρεπε ε, να πληρώσουν βαρύ ε, πρόστιμο για το θέμα αυτό οι χώρες μεσαίου μεγέθους τώρα για τις θέσεις που κατανέμονται σύμφωνα με τα διεθνικά ψηφοδέλτια. Ποιος κερδίζει, ποιος χάνει. Τα ψηφοδέλτια αυτά αφαιρούν, αφαιρούν ισχύ από τα κόμματα και από τους πολίτες στα κράτη-μέλη και δίνουν ακριβώς αυτή την ισχύ σε όσους ήδη στην Ευρωπή, στα ευρωπαϊκά κόμματα είναι ισχυροί σε αυτούς που αποφασίζουν ποιος θα είναι επικεφαλής ενός τέτοιου είδους ευρωπαϊκού ψηφοδελτίου. Αυτό θα είναι το αποτέλεσμα να αφαιρέσουμε δύναμη από τα χέρια των πολιτών και να την αποδώσουμε στους επικεφαλείς των ευρωπαϊκών κομμάτων. Πολύ κακή ιδέα αυτή. Αλλά βέβαια δεν σταματάει εκεί το θέμα. Έχουμε πρόβλημα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάποιες εθνικές αντιπροσωπείες είναι πιο ισχύρες. Αφήνοντας την άκρη ότι έχουν περισσότερα μέλη, αφήνοντας στην άκρη το γεγονός πως έχουν υπερεκπροσωπηθεί στις ανώτατες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλώ βέβαια για την ε, Γερμανία που είναι επικεφαλής ομάδων ευρωπαϊκών κομμάτων, ε, επιτροπών, υπερεκπροσώπηση. Και αυτό έχει να κάνει με την κρίσιμη μάζα των Γερμανών που μπορούν να μοιραστούν αρμοδιότητες, κάτι το οποίο δεν μπορείς να κάνεις όταν είσαι μικρή αντιπροσωπεία, μικρή χώρα. Έχουν λοιπόν περισσότερη ισχύ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και δεν νομίζω πως υπάρχει οποιοδήποτε στην αίθουσα αυτή που θα δείξει την παραμικρή έκθεση, την παραμικρή έκπληξη, αν σε περίπτωση διασυνοριακού ψηφοδελτίου ε, επικεφαλής και στις πρώτες θέσεις θα είναι άτομα από κράτη κράτη-μέλη τα οποία υπερεκπροσωπούνται. Οπότε αυτό είναι καλό η επιχείρημα κατά της χρήσης αυτών και κυρίως εδώ. Σας παρακαλώ πολύ συνάδελφοι να σέβεσαι το χρόνο. Δίνω το λόγο στη συνάδελφο. Ευχαριστώ λέει κυρία Μπρέσο. Δύο πράγματα να πω. Συμφωνούμε όσον αφορά την πρόταση της χρήσης με τους όρους που υπενθυμίστηκαν να χρησιμοποιήσουμε, λέγω, ένα μέρος των εδρών του Ηνωμένου Βασιλείου, εάν εξέρθει βέβαια να αποχωρήσει με μια ρήτρα που θα ισχύσει από τη στιγμή που επίσημα θα αποφασιστεί η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, ένα μέρος των εδρών να χρησιμοποιηθεί για να διορθωθεί η παρούσα κατάσταση και να σεβαστούμε αυστηρά την αρχή ε, της, της φθήνουσας αναλογικότητας. Δεύτερο θέμα. Η ομάδα μας συζήτησε τα υπερεθνικά ψηφοδέλτια και ήταν θετική. Σαν ομάδα εμείς είμαστε υπέρ των υπερεθνικών ψηφοδελτίων και πιστεύουμε ότι η πρόταση θα πρέπει να έχει συγκεκριμένα πλαίσια. Θα αξιολογήσουμε αν θα είναι δυνητική εφαρμογή αυτής το Κοινοβούλιο θα πρέπει να μπορεί να διαπραγματευτεί, να είναι έτοιμο να διαπραγματευτεί, αλλά η αφετηρία του Κοινοβουλίου πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι αυτή. Συνδέεται και με τον εκλογικό νόμο, κάτι που ζητήσαμε. Κάποιες θέσεις στο Συμβούλιο αλλάζουν πράγματι. Η Ιταλική κυβέρνηση ε, ήταν θετική, είναι θετική, θα είναι και η Γαλλική κυβέρνηση τώρα θετική. Αυτό μπορεί κάπως να κινήσει τα πράγματα. Βέβαια θα πρέπει εμείς να είμαστε διαθέσιμοι στις διαπραγματεύσεις να διαφοροποιήσουμε τις θέσεις μας. Αν είναι εφικτό όμως εντός του εκλογικού νόμου θα πρέπει να θεσπίσουμε κανόνες να είναι δημοκρατικό το εγχείρημα και να μην ενισχυθεί περαιτέρω η θέση των ισχυρότερων χωρών. Μπορούν να βρεθούν λύσεις για αυτά. Στο τελευταίο τμήμα. 27 θα είναι τα κράτη-μέλη σε αυτή τη φάση. Θα πρέπει ενδεχομένως να αφήσουμε σε αποθεματικό αν θέλετε κάποιο αριθμό εδρών για να χρησιμοποιηθούν σε κάποια μελλοντική διεύρυνση. Ευχαριστώ. Thank you, Ramon Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Χαουρέγγι για ένα λεπτό. Να πω πως το Κοινοβούλιο θα πρέπει οπωσδήποτε να καταθέσει μία πρόταση ε, ε βασιζόμενη σε μία μείωση εδρών ε, αφαιρώντας τις Βρετανικές έδρες. Αυτό θα πρέπει να γίνει έχει κοινοποιήσει το σχετικό άρθρο και εμείς αυτές τις 33 έδρες πρέπει να δούμε τι θα τις κάνουμε. Δεύτερον, εγώ είμαι υπέρ μιας πρότασης ενός διασυνοριακού διεθνικού ψηφοδελτίου και να σας πω ναι, χρειαζόμαστε αυτού του είδους το διεθνικό ψηφοδέλτιο γιατί πρέπει να κατανοήσουμε ποιο είναι το μήνυμα, ποιο είναι ο συμβολισμός για τον Ευρωπαίο πολίτη που θα ψηφίσει όχι μόνο ένα εθνικό ψηφοδέλτιο αλλά και ένα ευρωπαϊκό. Γιατί στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα έχουμε και κάποιους συμβολισμούς. Πάει κάποιο στην κάλπη όπου νομιμοποιείται το εκλογικό, μέσω εκλογικού σώματος η Ευρώπη, με τους 50-500 εκατομμύρια πολίτες, με ένα τέτοιο είδος ε, κοινό ψηφοδέλτιο. Είναι τεράστιος ο συμβολισμός, ακόμα και αν στην πράξη δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Και αυτά που είπε η Περβάρς, εντάξει, πρέπει κάπως να αντισταθμίσουμε ε, κάπως τις δυσκολίες που έχουν κράτη, οποία είτε λίγο απογραφής, είτε λίγο είτε κατανομής πληθυσμού, ε, που ε, πλήττονται ε, από τη σημερινή κατάσταση. Οπότε θα ήθελα να περιοριστούμε γύρω στις 725 έδρες στο Κοινοβούλιο για να καλύψουμε και αυτές τις ανησυχίες. Ραμόν, ευχαριστώ πολύ. Νομίζω πως τελειώσαμε. Δεν ξέρω αν Πέδρο είσαι απελπισμένος, απελπιστικά αναγκασμένος να ε, απαντήσεις, να σου δώσω το λόγο, ναι. Γι' αυτό τα ψηφοδέλτια να το ξανασυζητήσουμε. Είναι ένα θέμα το οποίο θα ξαναπροκύψει και θα πρέπει να αξιολογήσουμε τις διάφορες προτάσεις και να ξεχωρίσουμε και τα θέματα μεταξύ τους. Για το Brexit, επειδή γι' αυτό άκουσα κάποιες ε, ερωτήσεις, ναι, αναφέρθηκα σε μια μερική αναδιανομή των εδρών του Ηνωμένου Βασιλείου Αλλά αυτό το έκανα λαμβάνοντας υπόψη το χρονοδιάγραμμα του Brexit. Δηλαδή διατηρούμε το status quo μέχρι να τεθεί σε ισχύ το Brexit και μετά έχουμε μια νέα κατανομή εδρών η οποία μετά θα ισχύσει. Τώρα το πότε. Δεν έχω κάνει καμία αναφορά σε μεταβατική περίοδο. Ξέρουμε πως θα λάβει η χώρα το Brexit. Και ξέρουμε πως ε, όταν τεθεί σε εφαρμογή η συμφωνία αποχώρησης ή βέβαια μπορεί και μετά από δύο χρόνια και υπάρχει και ένα τρίτο σενάριο, μια ομόφωνη ε, απόφαση παράτασης. Οπότε νομικά υπάρχει κάποιο αβεβαιότητα. Σε πολιτικό επίπεδο η βεβαια μπορει και μετα απο δυο χρονια και υπαρχει ενα τριτο σεναριο μια ομοφωνη αποφαση παρατασης οποτε νομικα υπαρχει καποιο αβεβαιοτητα σε πολιτικο επιπεδο η ημερομηνια με την οποία αυτή τη στιγμή εργαζόμαστε είναι ο Μάρτιος του 2019 και γι' αυτό ως νομοθέτες πρέπει αυτή την ημερομηνία να τη λάβουμε δεόντως υπόψη προτάσεις μας. Το πρόβλημα είναι να είναι κανείς συνεισηγητής και πρόεδρος συνάμα. Νομίζω πως πρέπει να συνεχίσουμε. Ξέρω πως έχουμε και άλλα θέματα. Να σας πω μόνο πως ε, προσωπική μου άποψη και ξέρω πως Πέδρο έχετε και εσείς αυτή την άποψη πως εδώ είμαστε κοντά σε μια πλειοψηφία. Νομίζω σε σχέση με την κατεύθυνση που ακολουθούμε και ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχόλιά σας. Τα θεωρώ ιδιαίτερα υποστηρικτικά. Θέλω να σας ευχαριστήσω και νομίζω πως αυτό το οποίο έχουμε ετοιμάσει εμείς είναι μια κοινή κατανόηση των προκλήσεων που αντιμετωπίσει το Κοινοβούλιο τα επόμενα χρόνια. Μπορούμε λοιπόν Λοιπόν να μιλήσουμε για την πρώτη ανάγνωση το Σεπτέμβριο. 4 Σεπτεμβρίου λοιπόν και την πρώτη εργάσιμη μετά τις θερινές διακοπές θα λάβετε την έκθεση Κατόπιν θα συνεχίσουμε και νομίζω πως αν όλα πάνε καλά τον Νοέμβριο θα ψηφίσουμε στην Ολομέλεια. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον Πάολο Ράντζελ. Συμφωνήσαμε να μιλήσει σήμερα το πρωί γιατί έχει κάποια καθήκοντα που την καλούν στην Πορτογαλία το απόγευμα. 15 λεπτά. 15 λεπτά και δεν θα γίνει συζήτηση. Λυπάμαι πολύ. Έχεις το λόγο. Λοιπόν, είναι αρκετό γιατί Έχετε άλλωστε το έγγραφο για τις αποστολές αυτές, τις διερευνητικές, οι οποίες σχετίζονται και με την έκθεση που θα κάνουμε για την εφαρμογή των διατάξεων των συνδικών για τα Εθνικά Κοινοβούλια και για το θέμα αυτό θα ήθελα μόνο να υπογραμμίσω τρία ή τέσσερα σημεία, κάποιες ιδέες οι οποίες απορρέουν ως συμπεράσματα από τις δύο επισκέψεις που έκανα. Πήγα στη Δανία, στο Φόλκεντινκε τη Βουλή της Δανίας και επισκέφθηκα και την Ελληνική Βουλή. Επιλέξαμε το Κοινοβούλιο της Δανίας γιατί έχουν ένα μοντέλο εξέτασης μέσω εντολής οπότε θεωρείται το Κοινοβούλιο της Δανίας ε, ως ένα καλό παράδειγμα ε, της ε, εξέτασης των ευρωπαϊκών υποθέσεων και πήγαμε και στη Βουλή των Ελλήνων γιατί έχουν αυτό το πρόγραμμα διάσωσης και ήταν σημαντικό να δούμε πώς η Βουλή σε αυτά τα πλαίσια εξετάζει τα ευρωπαϊκά θέματα. Να σας πω πως αισθάνθηκα αρκετή έκπληξη γιατί και στις δύο περιπτώσεις άκουσα τις ίδιες απόψεις. Uh, rather interesting to see. Και ήταν αρκετά ενδιαφέρον το ότι οι Δανείοι βουλευτές, οι οποίοι έχουν τη φήμη πως είναι πολύ ισχυροί και έχουν πολύ ισχυρά δικαιώματα εξέτασης, ε, ε, κατήγγυλαν την κυβέρνησή τους. Και αυτό το οποίο διαπίστωσα και στην Κοπενχάγη και στην Αθήνα ήταν πως τα μέλη οι βουλευτές εξέφρασαν παράπονα για το επίπεδο ενημέρωσης από τις κυβερνήσεις. Και ήταν αρκετά ενδιαφέρον να διαπιστώνει κανείς πως πρόκειται για ένα γενικότερο, μια, ένα γενικότερο πρόβλημα το οποίο μοιράζονται και με τις ε, πολιτικές ομάδες της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Και στη Βουλή ε, των Ελλήνων ε, το αισθάνονται αυτό οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, όπως επίσης και οι ε, δανείοι βουλευτές κυβερνητικοί, οι οποίοι ήταν κατά της κυβέρνησή τους, γιατί θεωρούν πως όλες οι εθνικές κυβερνήσεις δεν παρέχουν επαρκή ενημέρωση εγώ αυτό φανταζόμουν πως μπορεί να συμβαίνει στη Βουλή των Ελλήνων, αλλά το γεγονός πως και οι Δανείοι, οι οποίοι συνήθως θεωρούνται πρότυπο, μια που έχουν αυτό το σύστημα εντολής και τα λοιπά, ε, εξέφρασαν ιδιαίτερη ε, δυσαρέσκεια με την κατάσταση και πρέπει να πω πως η κυβέρνηση της Δανίας ε, την τελευταία στιγμή ζητά την ε, την ε, έγκριση ε, της δικής τους βουλής, το οποίο σημαίνει ότι δεν μπορούν να επηρεάσουν τίποτα γιατί όλα έχουν περάσει από διαπραγματεύσεις. Οπότε είναι μια ελάχιστη, ένα ελάχιστο περιθώριο εξέτασης μπορούν να ασκήσουν. Αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα λοιπόν μου είπαν και στη Δανία και στην Ελλάδα και ήταν παρόμοια τα ζητήματα και ήταν και παρόμοιες εξηγήσει που άκουσα από τους βουλευτές των δύο αυτών κοινοβουλίων. Το παράδοξο βέβαια ήταν και ίσως ε, στο σημείο αυτό θα πρέπει να σταθούμε πιο πολύ είναι πως κυρίως στη Δανία μου ζήτησαν να έχουν περισσότερο έλεγχο, άμεσο έλεγχο επί των ευρωπαϊκών θεσμών. Δηλαδή είναι ξεκάθαρο για μένα ότι του ενδιαφέρει πιο πολύ να ελέγχουν του ευρωπαϊκού θεσμού, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε κάποιο βαθμό, αλλά κυρίω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί δεν έχουν επαρκή ενημέρωση από πλευρά τη δική του κυβέρνηση για τα θέματα αυτά. Οπότε σε αυτό το ζήτημα προφανώ υπάρχει κάποιο σφάλμα γιατί θα φανταζόταν κανεί πώ αφού ελέγχουν την εθνική του κυβέρνηση και η εθνική κυβέρνηση φτάνει στο Συμβούλιο με εθνική θέση, ε, προφανώς η νομοθεσία που προετοιμάζουν ε, έχει την έγκριση ε, ουσιαστικά του κοινοβουλίου τους. Αλλά οι 23 συστάσεις που έχω από τη Δανία, της Δανία τη Βουλή της Δανίας αποδεικνύουν πως δεν τους ικανοποιεί το σύστημα και θα προτιμούσαν ένα σχήμα όπου θα μπορούσαν να εισάγουν τροπολογίες απευθείας στη δική μας ε, νομοθετική διαδικασία. Οπότε θα είχαμε ένα είδος ε, ε τρίτης ε, ε τρίτου ελεγκτικού επίπεδου, ε, δηλαδή πέραν της πράσινης και της κίτρινης κάρτας ή της κόκκινης κάρτας, να υπάρχει και μια δυνατότητα ελέγχου μόνο από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Τώρα, μπορούμε να περάσουμε και στο γεγονός της ε, κατάθεση νομοθετικών πρωτοβουλίων. Αυτό μπορούν να το κάνουν μέσω τη δική σου εθνική κυβέρνηση. Δηλαδή μπορούν να ζητήσουν την κυβέρνησή του να καταθέσει μια νομοθετική πρόταση. Αλλά εκεί αντιμετήσουν το εξή πρόβλημα. Δεν είναι ότι υπάρχει κάποια ε, έλλειψη εμπιστοσύνη έτσι ώστε να επιθυμούν να, εξετα... να, να ελέγξουν ήδη τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Όχι. Είναι ότι αισθάνονται πω οι δικέ του κυβερνήσει δεν του ενημερώνουν επαρκώ για τα ευρωπαϊκά θέματα. Κάτι το οποίο εμένα μου προξένησε πάρα πολύ μεγάλη έκπληξη γιατί μου το επιβεβαίωσαν όχι μόνο ε, τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά ή φιλελεύθεροι στη Δανία και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή των Ελλήνων. Μας είπαν ότι και οι δύο ότι δεν μας ικανοποιεί καθόλου η δράση της κυβέρνησης εδώ. Τώρα, έχουμε και ένα άλλο θέμα, δύο άλλα θέματα στα οποία θα ήθελα να αναφερθώ και μετά θα κλείσω. Πρώτα απ' όλα να σας πω και αυτό θα το δείτε και στην έκθεση, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον να δείτε πόσο πολύ έχει προχωρήσει το σύστημα IPEX και πόσο καλά το λειτουργούν. Και εδώ μιλώ περισσότερο για τη Βουλή των Ελλήνων, η οποία συμμετέχει ιδιαίτερα με πολλές προτάσεις που τους επιτρέπουν να ανταλλάσσουν πληροφορίες και να κάνουν την εξέταση που χρειάζεται στο επίπεδο που προσφέρεται. Οπότε θα ζητήσουμε ε, να μας βοηθήσουν ε, ε, εμπειρογνώμονες από εκεί που έχουν για το IPEX γιατί πραγματικά ήταν εξαιρετικές οι ιδέες τους και έχουν ένα πολύ καλό τρόπο που λειτουργούν το όλο σύστημα. Επίσης, με πολύ ενδιαφέρον είδαμε πως η αξιολόγηση που κάνει η ΚΟΖΑΚ είναι τελείω διαφορετική από την κατάσταση α, την οποία διαπιστώσαμε πριν από 3-4 χρόνια. Δηλαδή, όλοι όταν μιλάνε για την ΚΟΖΑΚ λένε πω σήμερα λειτουργεί πολύ πιο επικοδομητικά, πω αποτελεί μια πλατφόρμα έτσι ώστε να δημιουργούνται καλές σχέσει μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Εθνικών Κοινοβουλίων. Αυτό έχει αλλάξει. Εγώ πρέπει να σα πω ότι έχω πάει σε πολλέ συναντήσει τη ΚΟΖΑΚ και ήταν πραγματικά χάλια. Δηλαδή, με συνεχή πίεση Πώς ε, κάνουν οι μαθητές όταν πάνε σχολείο και σε πιέζουν να κάνεις κάτι. Τέλος πάντων αυτό άλλαξε. Και λένε πως η Κόσακ πάει πραγματικά πολύ καλά. Και τέλος κάτι το πάρα πολύ ευαίσθητο και είναι η τελευταία πρόταση που θα πω. Και νομίζω έχουν δίκιο. Ανισχούν πάρα πολύ γιατί έχουμε την προθεσμία των 8 εβδομάδων για την ε, κίτρινη, για την πορτοκαλιά κάρτα, η οποία είναι υπερβολικά σύντομη. Αυτή η ιδέα που θα παρουσιάσω είναι δική μου, αλλά θα το δω με την νομική υπηρεσία. Θα προσπαθήσω να δημιουργήσω ένα σύστημα χωρίς να αλλάξω την νομοθεσία, ένα τεχνικό διάλειμμα πριν αρχίσουν να τρέχουν οκτώ εβδομάδες έτσι ώστε να παρατείνουμε ε, κατά 4 εβδομάδες αλλά ως τεχνική προετοιμασία. Ήταν πολύ ανοιχτή σε αυτή την πρόταση και κυρίως επειδή των ε, εξελίξεων που έχουμε και την πρόοδο στο IPEX δηλαδή να έχουμε αυτή την επιπλέον προθεσμία στο μέλλον. Τώρα, επειδή χάνω τη φωνή μου, θα πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, κοιτάξτε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ Περιμένουμε την έκθεσή σας. το Σεπτέμβριο θα συζητήσουμε την έκθεσή σας. Ελπίζουμε να μην αναβληθεί. Να προσθέσω κάτι. Αναφερθήκατε στην ΚΟΣΑΚ ότι προδεύει άριστα τα τελευταία χρόνια. Να σας πω ότι θα πρέπει και εμείς να επενεθούμε κάπως γι' αυτό. Και εγώ προσωπικά, αλλά με την ΑΦΚΟ τα τελευταία χρόνια έχουμε επενδύσει στην ΚΟΣΑΚ, υποστηρίξαμε κάποιε εξελίξει και συνεργαστήκαμε στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτω ώστε η ΚΟΣΑΚ να γίνει πιο επικοδομητική στο έργο τη. Άρα και ε, εμεί αξίζουμε κάποιον επένα. Πάμε στο σημείο 7 τη ημερήσια διάταξη. Έλεγα ότι μπορούμε να συζητήσουμε τώρα. Ε, Περβάνς θα διεξαχθεί συζήτηση το Σεπτέμβριο, διότι έχουμε μείνει πίσω, έχουμε καθυστερήσει. Δεν θα είσαστε. Α, θα είσαστε. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω, θα μιλήσετε για τον κύριο Φάβιο Καστάλτο για τους καταγγέλτες που ενεργούν προς το δημόσιο συμφέρον όταν αποκαλύπτουν πιστευτικές πληροφορίες επιχείρησης δημοσίων οργανισμών. Έχουμε γνωμοδότηση για την έκθεση ιδίας πρωτοβουλία, της Νομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Μπορείτε να είστε και εσείς σας παρακαλώ σύντομα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, όπως είπε και η Πρόεδρος, βρίσκομαι εδώ αντικαθιστώντας τον συνάδελφο Καστάλντο να σας παρουσιάσω την γνωμοδότηση για την έκθεση για τα μέτρα προστασίας ε, των καταγγελτών. Ο συνάδελφος Καστάλτο ζητά συγγνώμη, δεν μπόρεσε να είναι παρόν, διότι έχει ανελημμένες υποχρεώσεις για το Κοινοβούλιο σε μια συνάντηση στο Young Leaders Forum. Λοιπόν, να σα κάνω την παρουσίαση των θέσεων των. Όπω ήδη συζητήθηκε και αναφέρθηκε από την Πρόεδρο, το θέμα τη προστασία των ε, καταγγελτών είναι κρισίμου σημασία, κυρίω στην καταπολέμηση τη διαφθορά που ε, κοστίζει στην Ευρώπη περίπου 218 με 282 ε, δισεκατομμύρια ευρώ. Σε περίοδο μεγάλης ε, τέτοιας οικονομικής κρίσης πρέπει να το εξετάσουμε. Αυτοί οι καταγγέλτες είναι πολύ σημαντικοί για την καταπολέμηση της διαφθοράς και πρέπει να τους προστατεύσουμε. Ε, είναι ένα εργαλείο σημαντικό παρέμβασης. Είναι Λοιπόν, στο, κίνημα των πέντε αστέρων θεωρούμε ότι πρέπει να κινηθούμε σε την κατεύθυνση και κινούμεθα και σε εθνικό επίπεδο. Στα διαφορα κάτι κράτη-μέλη το θέμα αυτό αντιμετωπίζεται ποικιλοτρόπως και οι καταγγέλτε, δηλαδή πληροφοριοδότε, ε, την χάνουν κατακαιρματισμένη και τομεακή προστασία. Ε, λοιπόν, χρειάζεται μια ευρωπαϊκή κατεύθυνση ε, να είναι το πλαίσιο ευρύ και πλήρε. Και όσον αφορά ε, το επίπεδο της προστασίας και για τα θέματα για τα οποία προστατεύονται αυτά και ποιοι προστατεύονται. Βάσει αυτών εγώ ετοίμασα την γνωμοδότησή μου επικεντρωνόμενος επιθεσμικών θεμάτων και έτσι έχω κάποια σημαντικά σημεία. Όπως αναφέρεται στις συνθήκες, γίνεται σεβαστή δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση του κάτου δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Και η Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων προστατεύει πιο συγκεκριμένα μεταξύ άλλων και την ελευθερία της έκφρασης. Ε, μέχρι τώρα η παρέμβαση της ε, Ένωσης για την πράσπιση των πληροφοριδοτών όμως γίνονται στο μειακό επίπεδο και αυτό το λόγο ζητώ να εθετηθεί μια προπτική δράσεων ολιστική και οριζόντια. Ε, η συζήτηση επί του ουσίας για την νομική βάση που θα είναι δεδειγμένη είναι πολυπίκυλη. Στη γνωμοδότηση που συνέταξα Ζητείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αφού διεξαχθεί μια μελέτη συγκριτική των βελτίστων πρακτικών για το θέμα, να υιοθετήσει μια νομική βάση που θα εγγυάται την έγκριση ε, κοινού νομοθετικού πλαισίου σε τα κράτη-μέλη ε, και που θα είναι και το ευρύτερο δυνατό. Αυτό το νομοθετικό πλαίσιο θα πρέπει να καλύπτει και το δημόσιο τομέα και τον ιδιωτικό τομέα και να προστατεύει οποιονδήποτε αποκαλύπτει και εφιστά την προσοχή επιπληροφοριών για συγκεκριμένα γεγονότα. Το Συμβούλιο της Ευρώπης, ο ΙΕ και το Ευρωκοινοβούλιο επανειλημμένα υπογράμμισαν την πολύτιμη δημόσια λειτουργία προς όφελος όλων των πληροφοριδοτών. Ε, Παρ' όλα αυτά, αυτοί εξακολουθούν πολύ συχνά θύματα ε, στο να χάνουν τη θέση εργασία τους ή να αποκλείονται κοινωνικά και πολύ συχνά επεκτείνεται και στα μέλη τη οικογένεια τους αυτή η συμπεριφορά. Είναι σημαντικό λοιπόν οι πληροφοριδότε να προστατεύονται εγγυόμενοι ε, την μεγαλύτερη δυνατή ε, προστασία και θα πρέπει να προβλέπονται και μέτρα διαφύλαξης της φυσικής, ψυχολογικής και οικονομικής τους ακεραιότητας θα πρέπει να αλλάξει η κοινωνική αντίληψη αυτών των ανθρώπων διότι προσφέρουν σημαντική ε, ε, εξυπηρέτηση στην κοινωνία αλλά πολύ συχνά στιγματίζονται αρνητικά. Σχετικά με αυτό η τροποποίηση της πολιτισμικής προσεγγίσεως στο θέμα περνά και μέσω των ασφαλών διάβλων καταγγελιών που δίνουν ασφάλεια όσον αφορά την αντιμετώπιση των πληροφοριωτών από τη στιγμή θα κάνουν την καταγγελία τους και θα πρέπει να καλέσουμε τα κράτη-μέλη να προσπαθήσουν ενεργά να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Προτείνω λοιπόν να δημιουργηθεί ένα θέμα, μια ανεξάρτητη αρχή για την προστασία των πληροφοριοδοτών σύμφωνα ε, με την αρχή που εγγυάται την προστασία της ιδιωτικής ζωής. Θα πρέπει να αλλάξει το βήμα και η προσέγγιση. Από πλευρά των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων θα πρέπει να εφαρμόσουν πλήρω εσωτερικά ε, και ένα καθεστώς προστασίας και των υπαλλήλων που είναι προφοδότες και θα πρέπει να κάνει συστάσεις και ο διαμεσολαβητής Ευρωπαίος. Τέλος, σύμφωνα με την προαναφερθήσα προσέγγιση, πιστεύω ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία ισχύουσα θα πρέπει να εφαρμόζεται και από τους θεσμούς της Ένωσης και από τα κράτη-μέλη, ερμηνεύοντας με πιο θετικό τρόπο τα μέτρα για την προστασία των πληροφοριοδοτών. Αυτό συνοπτικά είναι το πλαίσιο της γνωμοδότησης που ετοίμασα και θα συμπεριλάβω και τις διάφορες ε, προτάσεις σας και ε, τροπολογίες για να είναι πληρέστερο το κείμενο. Η Νομική Επιτροπή ζητά την έγκριση της νομοδοτήσεως σε πολύ σύντομα. Η θα ψηφιστεί στις 28 Σεπτεμβρίου και θα πρέπει η γνωμοδότηση να τύχει μεγαλύτερη υποστήριξη. Θα πρέπει να διοργανώσουμε τουλάχιστον μια συνεδρίαση με του κοιόδη ηγητέ. Θα παρακαλούσα τη Γραμματεία να καθορίσει την ψηφορία τη γνωμοδοτήσεω κατά μια έκτακτη συνεδρίαση που θα λάβει χώρα κατά την Ολομέλεια του Σεπτεμβρίου στο Στρασβούργο. Και εσά, αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ υποβάλλετε τροπολογίε στα ελληνικά μέχρι τι 21 Ιουλίου. Ε, αναμονή τη συνεισφορά σα και είμαι βέβαιο ότι ε, θα είναι καρποφόρα η συνεργασία μα Αυτά και σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε δύο σκιώδεις εισηγητές που θα αναλάβουν το λόγο. Σας παρακαλώ να είστε πειθαρχημένοι στο βαθμό του δυνατού. Ραμόν, θα ήθελες να πεις κάτι σαν σκιώδης εισηγητής. Να πω μόνο πως θα παρουσιάσουμε τις αντίστοιχες τροπολογίες και είναι πιθανό να έχουμε και νομικά προβλήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή προσπαθώντας να βρούμε μια κοινή βάση. Πιστεύω πως δυστυχώς το σύστημα αυτό δεν μας δίνει αρκετές αρμοδιότητες, αλλά νομίζω ότι τα όσα είπε εκ μέρους του κυρίου Καστάλντου η συνάδελφος ε, θα βρουν την εξή ε, απάντηση. Νομίζω πως θα πρέπει να εξηγήσουμε πως αυτό το οποίο προσπαθούμε να προασπίσουμε εδώ είναι το δημόσιο συμφέρον. Δεν θέλουμε απλώς να τους προστατεύσουμε, αλλά θέλουμε να ενθαρρύνουμε κιόλας. Δηλαδή και νομίζω ότι στη Βόρεια Αμερική έχουν κάνει κάτι αντίστοιχο. Θέλουμε να δώσουμε κάποια κίνητρα έτσι ώστε οι υπάλληλοι να συμμετέχουν σε αυτές τις ε, καταγγελίες της ε, κακοδιαχείρισης, της ε, μη ικανοποιητικής λειτουργίας, ακόμα και της διαφθοράς. Και αυτό προσπαθούμε να το κάνουμε και μέσω της Επιτροπής Πάνα. Εκεί έχουμε το κεφάλαιο κατά της φοροπαφυγής και της φοροδιαφυγής, που είναι ουσιαστικά ζητήματα τα οποία οδηγούν και στις τις ε, παρουσιάσεις που ακούστηκαν και νομίζω πως τη γνωμοδότηση της ΑΦΚΟ θα την εμπλουτίσουμε με τις τροπολογίες που θα καταθέσει η ομάδα μας. Ευχαριστώ. Άντε και μετά Άντερσον. Ευχαριστώ πολύ. Θα θέλαμε και εμείς να σας ευχαριστήσουμε να ευχαριστήσουμε και τον εισηγητή για τις προσπάθειες που έκανε, για τις ιδέες του και να σας πω πως ε, συμφωνούμε πως οι, οι βάσεις, οι νομικές βάσεις είναι αδύναμες και θα πρέπει να προχωρήσουμε προσεκτικά γιατί ένα κομμάτι από αυτές τις αξιόπινες πράξεις που αποκαλύπτονται χάρη στους κατακέλοντες είναι διασυνοριακές από τη φύση τους. Οπότε θα πρέπει να μπορούμε να αποφύγουμε την ατιμορρησία με αυτή την άποψη το λέω και για να καταφέρουμε κάτι τέτοιο θα πρέπει να προκρίνουμε και να προστατεύσουμε όσο μπορούμε και με ό,τι μπορούμε εμείς να κάνουμε ε, τέτοιου είδους ε, καταγγελίες γιατί βέβαια υπάρχει ε, και το θέμα του κατά πόσο είναι χρήσιμες αυτές γενικότερα για την κοινωνία. Τώρα θα συνεργαστούμε επικοδομητικά με όλους τους συναδέλφους και είναι ένα θέμα που μας απασχολεί όλους ε, στην Πάνα, στη Λίμπε. Βλέπουμε πως η κοινή γνώμη το παρακολουθεί. Άρα λοιπόν θα πρέπει να προχωρήσουμε όσο μπορούμε πιο πολύ και να δούμε πώς μπορούμε να εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια που έχουμε. Ευχαριστώ για τους Ο Μαξ Άντερσον. Ελπίζω και εσείς να είσαστε όσο πειθαρχημένος ήταν συνάδελφοί σας. Ευχαριστώ. Πέντε σημεία έχω. Και θα τα αναφέρω ακροθυγός και σαφώς. Πρώτα, χρειάζεται οριζόντια προσέγγιση για την προστασία των πληροφοριοδοτών και όχι τομεακή. Γιατί? Διότι ο πληροφοριοδότης πρέπει να γνωρίζει ότι υπάρχει προστασία. Αν ακολουθήσουμε τομεακή προσέγγιση θα ποικίλουν κατά τομέα οι κανόνες, οπότε θα είναι πιο δύσκολο να είναι κάποιος πληροφοριοδότης. Δεύτερον, πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να προστατεύονται ανώνυμοι πληροφοριοδότες. Είναι εκείνοι που είναι κατά της ανωνυμίας, δοθέντος όμως ότι οι πληροφοριοδότες παρενοχλούνται πολύ συχνά, θα πρέπει να προστατεύεται και ο ανώνυμος πληροφοριοδότης, η ανωνυμία του πληροφοριοδότη. Μετά, στο άλλο σημείο, πράγματι σημαντικό να υπάρχει προστασία για την αντιμετώπιση της διαφθοράς στην Ένωση, αλλά πρέπει να πούμε κάτι και για τις λανθασμένες πράξεις. Υπάρχει επιθετικός σχεδιασμός φορολογικός, πράγματος χάρη, που δεν είναι κάτι παράνομο, αλλά πρέπει οι πληροφοριοδότες να μας βοηθούν να ξετρυπώνουμε τέτοια νομοθεσία και τέτοια μέτρα. Χρειάζονται κάποιες παράγραφοι για την προστασία των πληροφοριοδοτών Βεβαίως οι πράσινοι θα υποβάλουν σχετική τροπολογία για κεντρική ευρωπαϊκή αρχή βάση των εθνικών φορέων για την προστασία της ιδιωτικής ζωής. Δεν έχω πιστεί ότι κάτι τέτοιο είναι καλή ιδέα και προσβλέπω συνεδρίαση των σκιωδών όπου μπορούμε να το συζητήσουμε εκτενέστερα αυτό. Τέλος, οι πράσινοι θα προτείνουν τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Ταμείου για την προστασία των πληροφοριδοτών εκεί μπορεί να ζητήσουν νομική αρρωγή, ε, ψυχολογική στήριξη και να ζητήσουν αποζημίωση για παρενόχληση. Ευχαριστώ πολύ. Ο Τζορτ Σέφλιν για ένα ίσως ενάμιση λεπτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Από την Κωνσταντ Λεγκρίπ ανέλαβα το θέμα αυτό διότι έχει ε, κλεγεί, έχει έδρα στην Εθνική Γαλλική Εθνοσυνέλευση. Εντάξει, σας απαντήσω αυτό που είπατε. Κοιτάξτε, είναι χρησιμότατη αυτή η έκθεση. Οι πληροφοριοδότητες θα πρέπει να προστατεύονται. Πρέπει να προσέξουμε κάτι όμως. Υποτίθεται εν γέννη στην έκθεση και στα περισσότερα από αυτά που είπαν οι συνάδελφοι ότι είναι θετική η προσέγγιση όλων των πληροφοριοδοτών. Εγώ δεν πιστεύω ότι γενικά ισχύει. Μπορεί να είναι κακόβουλο το κίνητρο του πληροφοριοδότη. Μπορεί να φαίνεται ότι πρόκειται περί καταγγελίας, αλλά ίσως να αποκαλύπτει και εμπορικά μυστικά ο πληροφοριοδότης. Ίσως να προσπαθεί να καλύψει κατασκοπία. Υπάρχουν διάφορες πιθανότητες. Αυτό που λέω είναι ότι χρειαζόμαστε κάποιους όρους που πρέπει να θέσουμε. Πάνω απ' όλα η έκθεση θα πρέπει να λέει καθαρά ότι ισχύει μόνο για τον τομέα των εγκληματικών ποινικών πράξεων. Συγγνώμη, σας κάτσε για το τέλος, δεν ήξερα ότι σας η εισηγητής. Το αποφασίσαμε χτες. Εντάξει κύριε Πρόεδρε, δεν πειράζει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να πει κάτι. Όχι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Αντινόλφη θέλει να πει κάτι μήπως. Θέλετε. Κοιτάξτε, ε, κράτησα σημειώσει θα διαβάσω στον Φάβιο Μάσιμο Καστάλτο τις παρατηρήσεις και ελπίζω μετά να μπορέσετε ε, να συνεργαστείτε καρποφόρα. Ευχαριστώ. Πράγματι έχουμε χρονική πίεση. ψηφοφορία στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών και στην ΕΙΚΟΝ θα λάβει χώρα τέλος Σεπτεμβρίου. Θα πρέπει να έχουμε συνεδρίσει των σκιωδών τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου και ψηφοφορία στην Επιτροπή μας 4 Σεπτεμβρίου. Προθεσμία για υποβολή τροπολογιών είναι 20 Ιουλίου. Όσοι ενδιαφέρεστε, την 5η 20 Ιουλίου και θα προτιμούσαμε στα αγγλικά, παρακαλούμε στα αγγλικά, γιατί είναι δύσκολη η περίοδος του έτους, δεν έχω την ώρα. Ποιο είναι το χρονικό όριο. Τέλος της ημέρας. 5 λοιπόν το απόγευμα στις 20 Ιουλίου. Οπότε ολοκληρώνεται αυτό το σημείο. Να περάσουμε λοιπόν στο σημείο 8 της ημερήσιας διάταξης. Είναι η αποχώρηση του Ρωμαίου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις ανακοινώσεις ε, της Προέδρου δεν αναφέρθηκα στις τελευταίες εξελίξεις ε, του Brexit ε, γιατί έχουμε παρόντα εδώ τον Γκίφερ Χόφστατ ο οποίος είναι ο εκπρόσωπος του Κοινοβουλίου και ε, να σας δώσω το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Την προηγούμενη φορά που έκανα παρουσίαση στην Επιτροπή σας οι διαπραγματεύσεις δεν είχαν ξεκινήσει. Αλλά ούτε τώρα έχουν ξεκινήσει. Πολιτικά οι διαπραγματεύσεις θα ξεκινήσουν την ερχόμενη Δευτέρα. Οπότε θα έχουμε τον πρώτο γύρο των πολιτικών διαπραγματεύσεων τον οποίων προπαρασκευάζουν την τρέχουσα εβδομάδα ομάδες εργασίες και προβλέπονται τουλάχιστον τέσσερις ημέρες την επόμενη εβδομάδα τα θέματα αυτού του πρώτου γύρου θα είναι τρεις δέσμες θεμάτων. Πρώτη, δικαιώματα των πολιτών και θα επανέλθω αμέσως. Δεύτερον, λογαριασμός. Και ο τρίτος ε, αφορά ορισμένα και χωρισμένα θέματα. και σας τα λέω γρήγορα πυρηνικά θέματα και ασφάλεια των πυρηνικών καταστάσεων έχει να κάνει με την ε, Ευρατόμ τα προϊόντα που τίθεται στην αγορά διακυβέρνηση οι συνεχιζόμενες νομικές και διοικητικές διαδικασίες συνεργασία για αστικά και εμπορικά θέματα συνεχιζόμενη αστυνομική και ε, δικαστική συνεργασία για ποινικά θέματα και επίσης λειτουργία των θεσμών, φορέων και αρχών. Είναι 7 χωριστά θέματα με βάση 7 κείμενα θέσεων τα οποία αποφάσισε ο κύριος Μπάγνιε, ο διαπραγματευτής της Ένωσης Τεχνικά αυτή η τρίτη ομάδα εργασία άρχισε να συζητά σήμερα, ε, αυτή τη βδομάδα και πολιτικά η συζήτηση θα ξεκινήσει την ερχόμενη Δευτέρα. Αυτά τα τρία θέματα είναι χωριστά βέβαια, όπως βλέπετε. Αυτό που λείπει βέβαια είναι το θέμα των συνόρων μεταξύ της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας και της ε, Βορείου Ιρλανδίας. Εδώ υπήρξε μια συμφωνία μεταξύ των διαπραγματευτών των δύο πλευρών είναι να υπάρξει απευθείας διάλογος για το Ιρλανδικό θέμα. Να μην περάσει από ομάδες εργασίας. Να υπάρξει πολιτικός διάλογος με, μεταξύ της Σαμπίν Ράιαν που είναι η αναπληρώτρια του κ. Μπαρνιέ και του προσώπου Όλι Ρόμπινς του Ηνωμένου Βασιλείου που είναι επικεφαλής του Υπουργείου που ασχολείται με τον Brexit. Το λέω αυτό για να μην δημιουργηθεί η εντύπωση ότι χάθηκε το θέμα αυτό. Όχι, δεν ε, χάθηκε. Αντίθετα. Θα είναι το τέταρτο θέμα. Είναι θέμα κεφαλαιόδου σημασίας. Όπως θα γνωρίζετε, η ομάδα για το Brexit αποτελείται από εκπροσώπους των ομάδων που στήριξαν το αρχικό ψήφισμα που ενέκρινε το Κοινοβούλιο που εγκρίθηκε με πολύ ευρία πλειοψηφία. Λειτουργεί λοιπόν ε, με κανονικό ρυθμό και έχει αντιδράσει σε όλα τα κείμενα προτάσεων που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το κείμενο λοιπόν για τα δικαιώματα των πολιτών, το κείμενο για το λογαριασμό, την οικονομική διευθέτηση, τα 7 κείμενα θέσεων για τα 7 διαφορετικά θέματα. Για όλα αυτά έχουμε δώσει την άποψή μας με βάση φυσικά το ψήφισμα που ενέκρινε η Ολομέλεια και η ομάδα για τον Brexit του Κοινοβουλίου αντέδρασε και στο πρώτο κείμενο θέσεων που εξέδωσαν οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου για τα δικαιώματα των πολιτών πριν από μερικές εβδομάδες. Ελπίζω όλοι να βρήκατε τα mail με το αντίγραφο αυτού του κειμένου του κειμένου που έχει τίτλο αποτίμηση της ομάδας για τον Brexit, για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου που διαμένουν στην Ένωση και της Ένωσης που διαμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Επί του κειμένου αυτού, μαζί με τις υπηρεσίες αποφασίσαμε ότι ήδη αυτή τη βδομάδα θα θέσουμε στον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μια συγκεκριμένη σελίδα όπου όλοι οι συνάδελφοι και τα όργανα του Κοινοβουλίου θα μπορούν να στέλνουν τα κείμενά τους. Θα υπάρχει λοιπόν ένα χωριστό κουτί για τα ψηφίσματα. Υπάρχει μόνο ένα βέβαια μέχρι στιγμής, αλλά θα υπάρξουν και άλλα. Ένα άλλο σημείο όπου θα βλέπετε τις αντιδράσεις του Κοινοβουλίου στα κείμενα θέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όλες τις ε, τοποθετήσεις επ' αυτών πριν ολοκληρωθεί το κείμενο αυτό και χρησιμοποιηθεί στις διαπραγματεύσεις σε ένα τρίτο κουτί θα μπορείτε εύκολα να βρείτε τις αντιδράσεις της ομάδας του Κοινοβουλίου για τον Brexit στα κείμενα θέσεων του Ηνωμένου Βασιλείου τώρα περιέχει μόνο ε, μία αντίδραση για τα δικαιώματα των πολιτών και ένα τέταρτο κουτί για τη λυπή πληροφόρηση. Αλλά νομίζω ότι είναι απόλυτα ουσιώδες και θα γίνει ήδη αυτή τη βδομάδα. Θα ενημερωθούν όλα τα μέλη για το πώς μπορούν να αποστείλουν κείμενα σε αυτό το, αυτή την ιστοσελίδα, ούτως ώστε όλοι οι συνάδελφοι να μπορούν να παρακολουθούν τα κείμενα τα οποία εκπονούμε. συμβάλλοντας στη συζήτηση με βάση τα κείμενα του κ. Μπαρνιέ, του Ηνωμένου Βασιλείου και επίσης τα δικά μας ψηφίσματα για να υπάρχει πλήρης διαφάνεια. Όχι από πλευρά της Επιτροπής μόνο, αλλά και από τη δική μας πλευρά για το, το τι κάνουμε και το τι είναι διαθέσιμο. αλλά επειδή μόνο αυτή τη βδομάδα ολοκληρώνεται αυτή η προσπάθεια από τις υπηρεσίε του Κοινοβουλίου, σας έστειλα ήδη το δικό μας κείμενο για τα δικαιώματα των πολιτών και θα το έχετε δει αυτό το κείμενο. Θα είναι το πρώτο κείμενο που θα τεθεί στις διαπραγματεύσεις. Είναι προτεραιότητα του Κοινοβουλίου βεβαίω επίσης για το, τους πρώτους αυτούς γύρους των διαπραγματεύσεων. Τα δικαιώματα των πολιτών δηλαδή. Θεωρούμε ότι η πρόταση του Ηνωμένου Βασιλείου, της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου, είναι απολύτως αντίθετη από αυτό που θα θέλαμε. Από εκεί που θα θέλαμε να καταλήξουμε κατά το πέρας των διαπραγματεύσεων. Και είναι εντελώς αντίθετο με τη δική μας πρόταση για τα δικαιώματα των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου, όπου προτείνουμε απλώς να διατηρηθούν τα δικαιώματα και το καθεστώς των ε, δύο πλευρών, των πολιτών Τη μια πλευρά που διαμένει στην άλλη. Δηλαδή να το κατοχυρώσουμε αυτό, να το διασφαλίσουμε. Ενώ η πρόταση του Ηνωμένου Βασιλείου δημιουργεί το λεγόμενο σταθερό καθεστώς, όπως το αναφέρουν, settled status, που βασίζεται σε πενταετή παραμονή στη χώρα, το οποίο πρέπει να το ζητήσει μεμονωμένα ο κάθε πολίτης, δηλαδή θα πρέπει να δημιουργηθούν εκατομμύρια διαδικασίε. Δεν αρκεί ανά είναι ανάτομο. Δηλαδή, αν έχει δύο παιδιά, είναι άλλε δύο αιτήσει που πρέπει να κάνεις. Επίσης, δεν σέβεται πλήρω τα δικαιώματα που έχουν αυτή τη στιγμή οι πολίτες της Ένωσης στη Βρετανία κυρίως για θέματα επανένωσης οικογενειών αλλά και για παράδειγμα τα δικαιώματα τα οποία έχουν τώρα συμμετοχής στις, εκλογές, στις τοπικές εκλογές θα καταργηθεί και επίσης δημιουργείται ένα μεγάλο γραφειοκρατικό βάρος και τίθεται το ερώτημα Θα πρέπει οι πολίτες της Ένωσης ε, στο μέλλον, εάν διαμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, να εκλοφορούν με διάφορα χαρτιά για να αποδεικνύουν ότι έχουν δικαίωμα να είναι στη χώρα. Ενώ τώρα δεν έχει κανεί τέτοιο χαρτί. Δεν υπάρχει ταυτότητα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ενώ οι πολίτε τη Ένωση θα πρέπει να έχουν χαρτιά. Και φυσικά προτείνουν να ελέγχονται όλα αυτά από το Βρετανικό δικαστικό σύστημα. Υπάρχουν και λεπτομέρειες, ε, δεν θα τις αναφέρω. Θα τις βρείτε στο τετρασέλιδο κείμενο που στείλαμε σε όλους τους συναδέλφους. Προχθές. Επίσης, όχι μόνο δημιουργεί πολίτες δεύτερης κατηγορίας για τους πολίτες της Ένωσης, αλλά είναι απόλυτα αναντίστοιχο με τα δικαιώματα των Βρετανών στην υπηρετική Ευρώπη. Και εμείς δεν θέλουμε να μειώσουμε τα δικαιώματα των Βρετανών πολιτών στην υπηρετική Ευρώπη. Θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι είναι πολύ δύσκολο να γίνει του η Ευρωπαϊκή Δημοκρατία δεν δημιουργήθηκε για να μειώνεται το επίπεδο των δικαιωμάτων. Πρέπει τουλάχιστον να τα διατηρεί. Άρα δεν θα το κάνουμε. Η πρότασή μας λοιπόν προς τον Μισελ Μπαγνιέ στην αρχή των διαπραγματεύσεων τη Δευτέρα, η πρόταση που θα γίνει λοιπόν την επόμενη Δευτέρα, θα είναι να γίνει εξίσωση προς τα πάνω. Να ζητήσει δηλαδή να αυξηθούν τα δικαιώματα των, πολιτών της Ένωσης στις Ένωσης και να μην γίνει καμία απόπειρα μείωσης των δικαιωμάτων των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου που διαμένουν στο υπόλοιπο της Ένωσης γιατί οι πολίτες δεν θα πρέπει να πληρώσουν τα σπασμένα αυτής της διαδικασίας και το δεύτερο πρόβλημα που έχουμε υπάρχει πολύ ασάφεια στις προτάσεις του Ηνωμένου Βασιλείου υπάρχει ασάφεια για την ημερομηνία διακοπής του ισχύοντος καθεστώτος για τα κριτήρια για να αποκτήσει κανείς αυτό το ειδικό σταθερό καθεστώς δεν αναφέρονται ορισμένε κατηγορίες πολιτών, για παράδειγμα διαμεθοριακοί εργαζόμενοι. Δεν αναφέρονται. Δεν ε, αναφέρεται τίποτα για την αναγνώριση των επαγγελματικών τίτλων. Και επίσης, κάτι που είναι πολύ σημαντικό για την ευρωπαϊκή πλευρά, δεν αναφέρονται οι σπουδαστές. Δεν αναφέρεται. Δεν μπορεί να υπάρχει αβεβαιότητα για τους σπουδαστές. Πρέπει να υπάρχει βεβαιότητα, γιατί κάθε χρόνο αρχίζει η πανεπιστημιακή χρονιά. Δεν πρέπει να υπάρχει ασάφεια για το τι θα γίνει μέχρι την ημερομηνία αποχώρησης. Και κάτι άλλο που επίσης το ανέφερα ήδη, δημιουργούνται πολύ βαριές γραφειοκρατικές διαδικασίες. Ή δηλαδή το παράδειγμα ότι πρέπει κάθε μέλος της οικογένειας να κάνει χωριστά αίτηση. Επίσης, ποιοι θα είναι οι μηχανισμοί εφαρμογής αυτών των μέτρων. Εάν το σύστημα αυτό λειτουργήσει μέσω της Βρετανικής Υπηρεσίας Μετανάστευσης, και της ε, Βρετανικής νομοθεσίας μόνο δεν είναι επαρκές. Πρέπει να βασιστεί σε μια διεθνή συμφωνία μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτω ώστε να υπάρχει αυτόματα και διαδικασία επιτήρησης από την πλευρά μας από το ΔΕΚ Αυτά λοιπόν αλλά πιο λεπτομεριακά την αντίδραση και τις παρατηρήσεις μας προς τον Μισελ θα τα βρείτε στο κείμενο. Και αύριο θα έχουμε την τελευταία συνάντηση του Μισελ με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το θέμα αυτό πριν την έναρξη των διαπραγματεύσεων την προσεχή Δευτέρα. Τώρα για την ε, οικονομική διευθέτηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι στιγμής δεν έχει λάβει γραπτή πρόταση από τον Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε καν αν το Ηνωμένο Βασίλειο αναγνωρίζει ότι πρέπει να υπάρξει κάποια οικονομική διευθέτηση. Αυτή η αβεβαιότητα πρέπει να διαλυθεί αμέσως μόλι ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις. Δεν μπορούμε να πούμε ε, να συζητήσουμε ένα θέμα για τα άλλα θέματα δεν ε, συμφωνούμε καν ότι τίθενται. Ε, είναι λίγο υπερβολικά πρόχειρη αυτή η κατάσταση. Θα πρέπει να λάβουμε τη στάση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την πρόταση που κάναμε για το κείμενο θέσεων για την οικονομική διευθέτηση. Δεν ισχύει και αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Τα κείμενα βέβαια για τα άλλα 7 θέματα ευρατών και τα λοιπά δεν ε, δημοσιεύτηκαν μάλλον πρόσφατα. Οπότε είναι φυσιολογικό να μην υπάρχει αντίδραση. Τώρα το θέμα της Ευρατόμ επίσης δημιούργησε πολλά ερωτηματικά τις τελευταίες μέρες. Εδώ δίνω μόνο την προσωπική μου γνώμη, γιατί η ομάδα του Κοινοβουλίου για τον Brexit θα συζητήσει το θέμα αυτό σε προσεχή συνεδρίαση. Όπως καταλαβαίνω εγώ τις συνθήκες, μετά την ε, συνθήκη της ε, Λισαβόνας, οι δύο συνθήκες, Λισαβόνα και Ευρατόμ, συνδέονται το Ευρατόμ ε, χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό, η επίβλεψη γίνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, άρα δεν μπορεί να ανοίξει στο ένα ή άλλο Αυτό που θα ήταν δυνατόν, και αυτό προτείνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι να υπάρξει μια συμφωνία σύνδεση. Αυτή είναι η πρότασή μα. Να υπάρξει μια συμφωνία σύνδεση με βάση το άρθρο 217, στην οποία μπορούν να τεθούν όλα αυτά τα θέματα. Μπορεί να υποβάλει αίτημα το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ευρατόμη να συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντα που ασκεί τώρα. Και μπορεί να γίνει και στο μέλλον, βέβαια, ε, με αντάλλαγμα μια πληρωμή, γιατί δεν υπάρχουν μόνο δικαιώματα, αλλά και υποχρεώσει. Αλλά αυτό θα πρέπει να ρυθμιστεί σε μια μελλοντική συμφωνία σύνδεση. Δεν είναι τώρα θέμα τη στιγμή. Δεν είναι δυνατόν να αποχωρήσει κανείς από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να παραμείνει πλήρες μέλος της Ευρατόμ. Ούτε το αντίστροφο βέβαια. Γιατί μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας, από τη συνθήκη της Λισαβόνας και μετά, και οι δύο συνθήκες είναι παραρτήματα της βασικής συνθήκης που είναι η συνθήκη της Λισαβόνας. Αλλά αυτή είναι η προσωπική μου ταπεινή γνώμη. Είναι σαφές όμως ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα. Πρέπει να διευθετηθεί. Και αυτό το αναγνωρίζουμε και εμείς στην αντίδρασή μας στο κείμενο Μπαρνιέ. Είπαμε ότι το κύριο μέλημά μας είναι ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να συνεχίσει να σέβεται τις ενωσιακές προδιαγραφές για την πυρηνική ασφάλεια, τα ραδιενεργά απόβλητα και την διάθεση των αποβλήτων και θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της, τις ευθύνες του το Ηνωμένο Βασίλειο, για θέματα επαιτειότητας. Αυτή είναι μια σαφή θέση που πήραμε ως ομάδα του Κοινοβουλίου για τον Brexit και τη στείλαμε στον κύριο Μπάρνιε. Για να δούμε λοιπόν ποια είναι τα επόμενα βήματα. Καταρχήν τη Δευτέρα ξεκινούν οι πολιτικές διαπραγματεύσεις. Θα γίνει ένα briefing μετά από μία εβδομάδα και ο επόμενος γύρος διαπραγματεύσεων προβλέπεται να γίνει η τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου και θα ακολουθηθεί και αυτό από ένα briefing, μια σειρά από briefing μετά. Η πρότασή μου είναι να επανέλθω τότε στην ΑΦΚΟ και κάποια στιγμή αρχές Σεπτεμβρίου να σας κάνω μια καινούρια παρουσίαση. Τώρα, για τις περαιτέρω εργασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πιστεύω πως ίσως χρειαστεί να προετοιμάσουμε ένα καινούριο ψήφισμα για την Ολομέλεια που θα λάβει χώρα αρχές Σεπτεμβρίου και εκεί να αντιμετωπίσουμε κάποιες εκκρεμότητες, κάποια κρίσιμα ζητήματα, για παράδειγμα για τα δικαιώματα πολιτών, τα οποία ε, απέφχομαι βέβαια να είναι ακόμα τότε σε ε, εκκριμότητα, αλλά να έχουμε τη δυνατότητα τότε να εκφραστούμε και να επαναλάβουμε με μεγαλύτερη ευκρίνεια τα όσα είπαμε στο πρώτο μας ψήφισμα αν χρειάζεται. Γιατί βέβαια καταρχήν πρέπει να αποφασίσουμε αν όντω κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο, αλλά να υπάρχει δυνατότητα. Και νομίζω πως εκείνη τη στιγμή θα ήταν και ζωτική σημασία να επαναλάβουμε τις ανησυχίε που έχουμε ε, για τη συμφωνία ε, της ε, Good Friday στην Βόρεια Ιρλανδία και για τα θέματα γενικότερα τη περιοχή αυτή και το πώ θα αντιμετωπιστούν. Γιατί υπάρχει αυτή η αβεβαιότητα και νομίζω ότι οι κοινότητες εκεί ανησυχούν ιδιαίτερα. Έχουν δημιουργεί τρεις ε, ε, ομάδες εργασίας και ξαφνικά είπαμε «Α, ναι, και τα σύνορα μεταξύ ε, Βορείου Ιρλανδίας και Δημοκρατίας Ιρλανδίας είναι ένα θέμα για τους αναπληρωτές, θα τα δουν ξεχωριστά». Υπάρχει μία βεβαιότητα και νομίζουμε ότι εμείς θα πρέπει να δώσουμε φωνή σε όσους ανησυχούν, να θίξουμε το θέμα και να υπογραμμίσουμε πως δεν μπορεί το ζήτημα αυτό να αντιμετωπιστεί ξεχωριστά, το οποίο αφήνουμε στην άκρη ε, στο μισοδιάστημα. Κάτι στο οποίο νομίζω έχω αναφερθεί προηγουμένως, θα πρέπει φαντάζομαι τον Οκτώβριο το Κοινοβούλιο να κάνει και μια αξιολόγηση. Δηλαδή, να αξιολογήσουμε το κατά πόσο έχει ε, σημειωθεί επαρκής πρόοδος έτσι ώστε να μπορούμε, ναι ή όχι, να περάσουμε στη δεύτερη φάση των διαπραγματεύσεων που είναι η μελλοντική μας σχέση. Γιατί γνωρίζετε και εσείς πως οι καθεστητήρες γραμμές που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβολίο λέει πως ναι, μπορούμε να ξεκινήσουμε πριν το επίσημο, την επίσημη η υπογραφή ε, της συμφωνίας υποχρέωσης στις διαπραγματεύσεις για τη μελλοντική σχέση εφόσον έχει σημειωθεί επαρκής πρόοδος. Άρα λοιπόν είναι τμήμα του ρόλου του Κοινοβουλίου να παρακολουθήσει και να εξετάσει κατά πόσο την κατάλληλη στιγμή έχει σημειωθεί αυτή η επαρκή πρόοδο και αυτό να το κάνουμε πριν λάβει την απόφαση τη σχετική το Συμβούλιο. Νομίζω αυτό είναι ο ρόλο μα, ο ρόλο του Κοινοβουλίου και νομίζω ότι αυτή τη δουλειά θα πρέπει να την ξεκινήσουμε μέσα στους επόμενους μήνες. Και πιο πιθανό είναι να γίνει κάτι τέτοιο τον Οκτώβριο. Αυτά είχα να πω ως ε, ενημέρωση και αν θέλετε τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, αν πιστεύετε ότι είναι δυνατό να ξαναέρθω στην ΑΦΚΟ στα πλαίσια του προγράμματος να σας κάνω κάτι αντίστοιχο. Ευχαριστώ πολύ εκεί ένα θέμα ίσως ε, δεν αναφέρατε, ότι όταν είμαστε ε, σε αυτή την ομάδα για το Brexit, ε, γιατί είμαι και εγώ μέλος, όταν έχουμε ζητήματα τα οποία είναι αρμοδιότητα συγκεκριμένων επιτροπών, καλούμε την Προεδρία αυτών των επιτροπών για να λάβουν το λόγο. Και κάτι ακόμα στο οποίο θα ήθελα να σταθώ και να προσθέσω ενδεχομένω το θέμα των συνόρων. Αυτό προκύπτει επιπλέον από το γεγονός πως θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις μελλοντικές διευθετήσεις, οπότε είναι πολύ δύσκολο τώρα να κρίνουμε. Πάντως σας ευχαριστώ, έχουμε δύο συναδέλφους οι οποίοι θέλουν να κάνουν ερώτηση και να κάνουν σχόλια, νομίζω είναι μάλιστα παραπάνω από δύο. Συνάδελφοι, έχουμε 20 λεπτά, Λάινεν, Σέπλιν, Κόλπρεκ, James. Κάποιος ακόμα. Οκ, Μέρι Μακίνες. Δεν σας βλέπω, σηκώστε το καρτελάκι σας. Πολύ ωραία. Νομίζω ότι και εδώ θα πρέπει να δείξουμε πολύ πειθαρχία. Α, μην κάνετε μακροσκελή σχόλια, ζήτηστε να σας απαντήσουν σε ερωτήσεις. Απευθύνετε τις ερωτήσεις σας στον ΚΙ. Και να σας πω πως στην διευθύνουσα αυτή ομάδα που έχουμε κυρίως εκπροσώπους πολιτικών ομάδων, αυτό που συμβαίνει είναι Κατά σύμπτωση να έχουμε τρία πλήρη μέλη της ε, Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων ε, και ένα αναπληρωματικό. Είμαι και εγώ, οπότε έχουμε μια εκπρόπηση. Ο κύριος Λάινεν έχει το λόγο. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Κίφερ Χόστατ για τη διαφάνεια την οποία επιδεικνύει, την οποία μας είχατε υποσχεθεί και την οποία εφαρμόζεται και στην πράξη γιατί βγάζετε όλα τα έγγραφα στο διαδίκτυο και νομίζω πως πολλοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουν να παρακολουθήσουν τι γίνεται με το πρώτο διαζύγιο ενός κράτους μέλους από την Ευρωπαϊκή Ένωση και βέβαια η διαφάνεια και τα έγγραφα είναι το πρώτο βήμα. Το πρώτο τεστ που θα περάσουμε είναι τα δικαιώματα των πολιτών, να δούμε αν εμείς είμαστε αξιόπιστοι, αν σεβαστούμε τις υποσχέσεις μας, αν τα κάνουμε όλα στον κατάλληλο χρόνο και βλέπουμε ήδη πως υπάρχει μια μεγάλη διαφορά των ε, δικαιωμάτων που απολαμβάνεις όταν είσαι πολίτης Ευρωπαϊκής Ένωσης και των δικαιωμάτων που έχεις απλώς ε, ε, το καθεστώς που έχει το Ηνωμένο Βασίλειο που προσπαθεί να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, και γι' αυτό θα πρέπει για τα 3 εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο να διατηρήσουμε στο βαθμό που μπορούμε το status quo και ίσως να έχουν ένα ξεχωριστό στάτου στο μέλλον, ένα ξεχωριστό καθεστώς ε, ως πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαβιώνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τώρα, για τα οικονομικά θέματα, χτες το βράδυ είχα πάει σε μια διάσκεψη για την ε, Ενεργειακή Ένωση, για τον Brexit και έμαθα πολλά για τη Euratom. Κανείς δεν γνωρίζει πως τα πυρηνικά υλικά και ο εξοπλισμός ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ουχή στα κράτη-μέλη. Το Sellafield ε, παράγει πάρα πολλά απόβλητα για τα, ε, που έρχονται στα κράτη-μέλη, οπότε νομίζω ότι το θέμα αυτό θα, θα δημιουργήσει προβλήματα. Ξέρω πως αυτή τη στιγμή ε, οικοδομούμε 10 βρόμχους από την υπηρετική Ευρώπη προς το Ηνωμένο Βασίλειο και η επένδυση είναι της τάξης των 9 δις ευρώ για υποδομές ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν, συγγνώμη, στο λογαριασμό εκαθάρισης αυτά τα 9 δις θα έχετε τοποθετήσει, γιατί εμείς αυτή τη στιγμή χάνουμε ενεργειακές υποδομές. Και επίση Τετάρτη απόγευμα, να σας πω, όχι, Δευτέρα απόγευμα, το Συμβούλιο Ενέργειας αποφάσιζε ποιο θα είναι το θεματολόγιο για το 2030, για την ενεργειακή αποδοτικότητα. Και συνάδελφοι μου είπαν πως το Ηνωμένο Βασίλειο έδειξε ιδιαίτερο ενθουσιασμό για να επηρεάσει τους στόχους για την ενεργειακή αποδοτικότητα και βέβαια καταφθάνουν συνέχεια ερωτήσεις για το ποιο είναι ο ρόλος ε, του Ηνωμένου Βασιλείου στην νομοθεσία που ξεπερνά τα χρονικά όρια του 2020. Ξέρω ότι υπάρχει πρόβλημα, αλλά θα πρέπει να το συζητήσει κανείς. Δηλαδή, μπορούν να επηρεάσουν άμεσα και τι θα κάνουμε εμείς αφού φύγουν. Έχουμε πολλούς ομιλητές, οπότε στα δύο λεπτά θα χτυπάει το σφυράκι. Για να μας απαντήσει και ο Γκίς ερωτήσεις μας ο Τζόρτζ Σέπφλιν. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ τον Γκίφερ Χόφστατ για αυτή την παρουσίαση που είναι εξαιρετικά χρήσιμη. Θα είμαι πολύ σύντομος. Νομική αβεβαιότητα και το σχετικό πρόβλημα. Νομίζω είναι κομβικό και γιατί υπάρχει το θέμα της εθνικής κυριαρχίας του, της ε, Βουλής ε, των Κοινοτήτων στο Westminster. Όλα μπορούν να καταργηθούν, έστω και αναδροματικά μπορούν να αποσυρθούν. Οπότε το λιγότερο που μπορούμε να ζητήσουμε είναι μια διεθνή ε, συμφωνία με έναν ανεξάρτητο μηχανισμό επίλυση διαφορών. Είναι έτοιμο το Ηνωμένο Βασίλειο. Γιατί ο λόγος για τον οποίο θέλουν να πάρουν πίσω τον έλεγχο είναι να εξασφαλίσουν την απόλυτη εθνική κυριαρχία των όσων κάνουν από το Westminster άλλο. Κάποιοι πολίτες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ηνωμένο Βασίλειο και χρησιμοποιώ την ορολογία ε, με απόλυτη συνείδηση είναι Ιρλανδοί πολίτε. Τι θα γίνει τώρα δεδομένης, δεδομένου και των συνόρων και των ειδικών σχέσεων μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Δημοκρατίας Ιρλανδίας. Ο κύριος Κόλμορ, τι πιστεύετε γιατί θα ήθελα και εγώ να σχολιάσω ε, για κάτι το οποίο για μένα αποτελεί βασική δυσκολία στις διαπραγματεύσεις αυτή τη στιγμή. Είναι τι πιστεύετε, υπάρχει αυτή η έλλειψη σαφήνειας για το ποια είναι η θέση του Ηνωμένου Βασιλείου. Για όλα σχεδόν τα σημεία κλειδιά. Η πρώτη συνάντηση στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων ήταν αξιοσημείωτη από το γεγονό πω δεν κατέθεσαν ούτε ένα έγγραφο θέσεων ούτε πριν ούτε κατά τη συνάντηση. Έκτοτε έχουν υποβάλει ένα, στο οποίο αναφερθήκατε, αλλά δεν έχουμε κανένα έγγραφο θέσεων για οποιοδήποτε από τα υπόλοιπα θέματα. Ίσως λόγω του χάους και της σύγχυσης που επικρατεί στη Βρετανική κυβέρνηση που ακόμα δεν γνωρίζει τι θα ζητήσει για πάρα πολλά από αυτά. Έχετε λάβει κάποιες ενδείξεις για πότε θα κατατεθούν ενδεχομένως κάποια από αυτά τα έγγραφα με την περιγραφή των θέσεων. Δεύτερον, δεδομένης της έλλειψη χρόνου που είναι εντονότερη από ό,τι αρχικά είχε προβλεφθεί και δεδομένου του μεγάλου αριθμού θεμάτων και τι δυσκολίε που έχει η Βρετανική κυβέρνηση να λάβει θέση για πολλά από αυτά. Δεν βλέπετε να υπάρχει κάποιο κίνδυνο ε, το διαζύγιο μέσω άρθρου 50 θα ασχοληθεί μόνο με το ελάχιστο των θεμάτων που χρειάζεται να αποφασιστούν πριν γίνει το Brexit και όλα τα υπόλοιπα θα τα αφήσει για, ένα επόμενο, για μια επόμενη συμφωνία πλαίσιο ε, με ε, διατήρηση στο εντωμεταξύ, στο μεσοδιάστημα του status quo. Γιατί ξέρω πως και η Βουλή η Βουλή των Κοινοτήτων και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και γι' αυτό ανησυχούμε εμεί, εξετάσουν τη συμφωνία αυτή αποχώρηση, θα την εξετάσουν χωρί να γνωρίσουν πώ θα αντιμετωπιστούν κάποια από τα κομβικά ζητήματα. Και θα μα πούνε μην ανησυχείτε, θα το δούμε αργότερα, όλα θα πάνε καλά. Αλλά στην πραγματικότητα, και έχουμε μια έκφραση στα αγγλικά, γουρούνι στο σακί θα αγοράσουμε μας ζητούν κάτι να δεχτούμε και εμείς και η Βουλή στην Αγγλία να υπογράψουμε κάτι το οποίο τελικά δεν θα περιγράφει τι θα γίνει για βασικά θέματα. Ναι, Κοιτάξτε, το ότι δεν έχουμε αυτά τα έγγραφα θέσεις ίσως έχει να κάνει με την ε, δέσμευση υπέρ της διαφάνειας που έχουν τις δύο πλευρές. Προφανώς δεν έχουν την αντίστοιχη δέσμευση με εμά στο ε, Ηνωμένο Βασίλειο. Κύριε Τανζάνς, ε, καταρχήν, 69% του βρετανικού πληθυσμού θέλει ακόμα να φύγει. Αυτό είναι πάνω από το 52% του δημοψηφίσματος και 82% ήταν ήτανε υπέρ του των δύο κομμάτων που, υπερα, που ήταν υπέρ του Brexit. Οπότε νομίζω ότι η οργάνωση όλων αυτών των θεμάτων είναι εξαιρετικά ετεροβαρής και εμείς γέρνουμε σαφέστατα προς μία πλευρά. Κοιτάξτε, Έλεγχο μετανάστευση. θέμα εθνική κυριαρχία. Το Ηνωμένο Βασίλειο είπε ποια είναι η θέση του και η έκθεση είναι δίκαιη. Και έχουμε την έκθεση τη Τερέζα Μέη για το τι είχαμε εκχωρήσει ω ε, κράτος μέλους Ευρωπαϊκή Ένωση και τι θα ανακτήσουμε. Και για τον κύριο Φερχόφστα, να του πω τα εξή. Καταρχήν, δεν χρειάζεται να είναι κανεί μέλλον τη Ευρωπαϊκή Ένωση για να είναι μέλο του Εράσμου. και αν έχετε σκοπό να διώξετε όλα τα μη κράτη-μέλη από το ωραία, να δούμε πώ θα το καταφέρετε, ενδιαφέρουσα θέση. Και πείτε μου μου στα πλαίσια της διαπραγμάτευσής σας. Το 25% 2 ε, ε, δις ε, δανείων από Ευρωπαίους φοιτητές που δεν πλήρωσαν, δεν αποπλήρωσαν τα φοιτητικά τους δάνεια. Να δω. Και ξέρετε ποιοι είναι οι χειρότεροι κακοπληρωτέκτ. Η Γερμανία και η Γαλλία. Αρχιτέκτονες του Ευρωπαϊκού Οικοδομήματος. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Πάρτον. Ευχαριστώ πολύ. Πολλά θα ήθελα να πω, αλλά επειδή έχουμε λίγο χρόνο θα περιοριστώ σε ένα θέμα. Καταρχήν να πω πως η ευρωπαϊκή κυβέρνηση έκανε μια πολύ γενναιόδορη προσφορά, πολύ λογική. Και τι άλλο θα είχε κάνει. Ε, βέβαια, ε, εξατομικευμένα. Δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή εμείς να έχουμε ταυτότητα στη Βρετανία. Δεν είμαστε αστυνομιβόμενο κράτος και νομίζω ότι μπορεί σε κάποιες χώρες να χρειάζεται να αποδείξεις ποιος είσαι. Ναι, σε κάποιες χώρες στην Ευρώπη συνέχεια πρέπει να έχει ταυτότητα μαζί. Αλλά το θέμα που θέλω να πω είναι η αμοιβαιότητα και η δικαιοσύνη. Γιατί ο κύριος Φερχόφστας μιλάει για αυτό στο έγγραφό του και εδώ έχουμε τα δικαιώματα των πολιτών. Λοιπόν, έχουμε μια τεράστια έλλειψη ισορροπία μεταξύ του αριθμού των ε, πολιτών του, ε, ε, ε, του Ηνωμένου Βασίλειου που ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 1,2 εκατομμύρια και έχουμε και 3,2 εκατομμύρια πολίτες Ευρωπαίου που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Λοιπόν, Για τα ε, προνοιακά επιδόματα να σας πω πως αυτή τη στιγμή έχουμε μια βραδευλεγή βόμβα κάτω από το Brexit που είναι αυτό το θέμα. Μιλάτε εσείς για το δικαίωμα των ε, παιδιών που δεν έχουν γεννηθεί ακόμα το 2019, όταν δηλαδή θα φύγουμε, να ε, έχουν και αυτοί το δικαίωμα να πληρώνονται τα προνοιακά τους επιδόματα στο εξωτερικό. Ε, συγγνώμη. 883.000 περίπου Πολωνοί ζουν ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο. 35.000 Βρετανοί ζουν στην Πολωνία. Συγγνώμη, στα πλαίσια τη αμοιβαιότητα και τη δικαιοσύνη, Τα άτομα που είναι εκεί και ζουν εκεί και έχουν σε δικαιώμα σε προνοιακά επιδόματα, σε επιδόματα στέγης, ε, σε περίθαλψη, σε όλα τα δικαιώματα. Ε, εντάξει, Πώ θα δούμε την αμοιβαιότητα, γιατί οι Βρετανοί στην Πολωνία δεν θα έχουν το δικαίωμα σε επίδομα στέγη και σε ε, ε, υπηρεσίε του ΕΣΥ, γιατί εκεί δεν έχουν τα ίδια που έχουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οπότε για ποια δικαιοσύνη μιλάμε. Δηλαδή, οι φορολογούμενοι στη Βρετανία που τόσο σκληρά δουλεύουν να πληρώνουν επιδόματα πολιτών που ακόμα δεν έχουν γεννηθεί όταν δεν μπορούν να λάβουν ε, την ίδια παροχή, κοινωνική παροχή ε, κάπου αλλού που ζουν γιατί δεν υπάρχει το αντίστοιχο επίδομα. Εγώ ζω σε μια τι πιο ε, φτωχέ γειτονιέ του Λονδίνου και τι θα πω εγώ ε, στου εκλογέ μου, ότι θα πρέπει ε, αιωνίω να πληρώνουν φόρου για ανθρώπου οι οποίοι δεν ζουν καν στο Ηνωμένο Βασίλειο και όταν δεν έχουν οι ίδιοι το αντίστοιχο δικαίωμα, αν επιλέξουν κάποια στιγμή να πάνε να ζήσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελπίζω να μην σα παρανόησα, αλλά η αμοιβαιότητα δεν εξαρτάται από το μέγεθο του πληθυσμού ή του προβλήματο, είναι μια αρχή. Αλλά θα το συζητήσουμε και αυτό στις απαντήσεις. Η κυρία Μακίνης. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον κύριο Χόφστατ για την ενημέρωση. Πράγματι ήταν ανοιχτό και συνάντησε διάφορες αντιπροσωπείς, διότι πολλοί τον επισκέπτονται. Ποιο είναι το πρόβλημα που έχω όσον αφορά το θέμα των συνόρων. Υπάρχει μεγάλη ευαισθησία όσον αφορά αυτό το θέμα. Πιστεύετε ότι από πλευρά Ηνωμένου Βασιλείου γίνεται κατανοητό ότι όταν αποσυρθεί από την ενιαία αγορά και την Τελωνιακή Ένωση ταυτόχρονα ότι υπάρχουν συνέπειες και ίσως θα μπορούσατε να σας αναφέρετε πιο ξεκάθαρα όπως έκανε ο Μισελ Μπαρνιέ. Εν τη αυτή περιπτώσει, αν αυτό ισχύει, ανταποκρίνεται στις δεσμεύσεις του Ηνωμένου Βασίλειου Βασίλειο. Να είναι αόρατο το σύνορο, να μην γίνει επιστροφή στο παρελθόν Σχολιάστε το αυτό σας παρακαλώ. Αυτή την εβδομάδα είχα μία αντιπροσωπεία που συναντήσατε κι εσείς. Δεν ήταν πολιτική. Ήταν επικεφαλής ε, διαφόρων ε, συμβουλίων δημοτικών ε, για τις δύο πλευρές των συνόρων που συνεργάζονται. Είναι καλό για τον κόσμο που κατοικεί και από τις δύο πλευρές των συνόρων, που είναι κάτι αόρατο σε αυτή τη φάση. Ανησυχούν θα συνεχίσει αυτή η κατάσταση στο μέλλον. Τέλος μπορούμε να κάνουμε κάτι, να βοηθήσουμε το Ηνωμένο Βασίλειο να καταλήξει σε κάποια σωστή θέση. Όλοι προσφυσόμαστε τα συμφέροντά μας. Υπάρχει κάτι μεγαλύτερο από όλους μας. Η ειρηνευτική διαδικασία που είναι άκρος έθραυστη σε αυτή τη φάση και η πολιτική κατάσταση στη Βόρεια Ιρλανδία. Ο λαός της Βόρειας Ιρλανδίας δεν εισακούεται, δεν έχει φωνή, δεν υπάρχει συνέλευση. Και εμείς υπέχουμε το καθήκον να διαβιβάζουμε τις ανησυχίες όλων των κοινοτήτων της Βόρειου Ιρλανδίας. Ευχαριστώ ο Χέλμουτ Σόλτ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον Κίφερ Χόφστατ για τη διαφάνεια που επέδειξε. Ε, ερωτήσεις. Έχουμε συνομιλήσει με αρκετού πολίτε του Ηνωμένου Βασιλείου και τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Και όπω λέγεται, τίποτα δεν έχει συμφωνηθεί μέχρι να συμφωνηθούν τα πάντα όσον αφορά τα δικαιώματα. Και γι' αυτό ανησυχούν. Ερώτηση. Είχατε τη δυνατότητα να καταλήξει σε κάποια συμφωνία για τη δικαιώματα των πολιτών και να, τα διοχα... να διαχωρίσετε τα δικαιώματα των πολιτών από τις άλλες πτυχές της συμφωνίας. Υπάρχουν και άλλα θέματα, όπως το θέμα των συνόρων και άλλα ευαίσθητα ζητήματα. Υπάρχει το συνέστημα, πρέπει να υπάρχει το συνέστημα ότι δεν απεμπολούμε τα δικαιώματα των πολιτών στις διαπραγματεύσεις. Κυρίως στην τελευταία φάση. Μετά Έχουμε τη στη Διεθνή Επιτροπή, την Επιτροπή Διεθνούς Εμπειρίου ζητήσαμε και την άποψη νομικής υπηρεσίας για τις μελλοντικές εμπορικές σχέσεις. Σημαίνει ότι ήδη πρέπει να καταλάβουμε οι διεθνείς συμφωνίες, όπως η ΣΥΤΑ, η Συμφωνία της Σιγκαπούρης και άλλοι, πώς συνδέονται με τον όγκο των πληρωμών στον τελωνιακό τομέα. Οι υποχρεώσεις πώς θα κατανεμηθούν που απορρέουν από διεθνείς συμφωνίες με τρίτες χώρες. Και ποιος ασχολείται με αυτό το ζήτημα. Έχετε απαντήσεις για αυτά. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ζωητόφσκι. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σύντομα, θέλω να τονίσω το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα πρέπει να έχουμε όλοι σαν στόχο την σύναψη μιας συμφωνίας που είναι υποφελής και για το Ηνωμένο Βασίλειο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να είμαστε πρέπει να είναι ανοιχτή η λειτουργία διαφανής της διευθύνουσας αυτής της ειδική Επιτροπής. Πρέπει να εκπροσωπούνται όλες οι απόψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πρέπει να προσέξουμε ποια δράση θα εφαρμόσουμε. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να αξιολογεί τις ε, διαπραγματεύσεις και όχι να τις διαμορφώνει. Και γι' αυτό με προβληματίζει ε, άλλο ένα ψήφισμα που θα προσπαθούσε να διαμορφώσει τις διαπραγματεύσεις ακόμα πριν αυτές οι διαπραγματεύσεις φτάσουν σε ένα πιο κρίσιμο στάδιο. Ε, συντομία γι' αυτό. Η διευθύνουσα αυτή ομάδα, η ειδική ομάδα, εργάζεται για τη διάσκεψη των Προέδρων και στη διάσκεψη των Προέδρων έχουμε εκπροσώπους όλων των πολιτικών ομάδων. Αυτό έχετε το υπόψη. Τελειώσαμε λοιπόν με τις ερωτήσεις. Ε, αν μπορείς δώσε απαντήσεις, πολύ σύντομα. Ετέθη το ερώτημα. Είναι η ειδική κατηγορία Ιρλανδοί πολίτες. Ναι, διότι είναι Ιρλανδοί, πρώτα απ' όλα. Και δεύτερον, διότι έχουν αυτό τον κοινό ε, χώρο ε, μετακίνησης και οι Βορειοερλανδοί πολίτες, 1,8 εκατομμύρια έχουν δυνατότητα Ιρλανδικού διαβατηρίου. Ναι, και αυτό πιο πέρα ε, και για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Αυτό δεν το βλέπει κανείς σαν πρόβλημα. Κυρία Μαγκίνες, για το ίδιο ζήτημα. Στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου Υπάρχει ένα κομμάτι που έχει τροποποιηθεί και αναφέρεται σε όλα τα μέρη της Συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής. Δεν είναι τυχαίο που είπαμε όλα τα συμβαλόμενα μέρη. Αν εξετάσει τη Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής υπάρχει σαφής εγγύηση. Τίποτα δεν μπορεί να συμβεί να εφαρμόσουν τα μέρη της συμφωνίας να κάνει κάτι ένα από τα μέρη που καταστρέφει τις ισορροπίες της συμφωνίας. Και είναι σαφές ότι η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ενιαία αγορά αυτομάτως δημιουργεί σκληρά σύνορα ένα νέο εμπόδιο που είναι αντίθετο προς τη Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής. Όταν λέμε όχι σκληρό σύνορο, ε, δεν είναι μόνο κακό διότι υπάρχει ένα σύνορο, αλλά διότι είναι αντίθετο με τα συμπεφωνημένα ε, της ε, Συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής. Και γι' αυτό Κυρία Μαγκίνες, πιστεύω ότι σε αυτή τη φάση, αν θεωρήσουμε ότι χρειάζεται συμπληρωματικό ψήφισμα, πρέπει να το επαναξετάσουμε το ζήτημα και να αναφέρεται αυτό το σημείο στο ψήφισμα, να το υπενθυμίσουμε αυτό. Ε, τούτου λεχθέντος για την ώρα. Δεν είδα κάποια πρόταση που να είναι ε, καλή, ούτως ώστε να επιλύει 100% το πρόβλημα υπάρχει σύνορο. Δεν μπορεί να γίνει ένα ελεγχόμενο σύνορο, ένα σκληρό το σιπίν σύνορο. Τι σημαίνει αυτό άραγε. Δεν υπήρχε σύνορο διότι όλοι ανήκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην ενιαία αγορά. Και το θέμα είναι πού θα τεθούν τα σύνορα, πού θα μπει αυτό το σύνορο. Θα είναι χερσαίο σύνορο, θαλάσσιο σύνορο. Υπάρχουν πολλές δυνατότητες, ε, διάφορα θέματα προς αξιολόγηση από τη στιγμή που θα δούμε συγκεκριμένες προτάσεις για αυτό το θέμα. Είναι σημαντικό λοιπόν πριν ε, ξεκινήσει το όλο εγχείρημα να επαναλάβουμε κάποιες βασικές αρχές ως κοινοβούλιο απευθυνόμενοι προς τους διαπραγματευόμενους. Πρέπει να ανάψουμε το τελικό πράσινο φως για τη συμφωνία αλλά για να είμαστε βέβαιοι για να μπορέσουμε να ανάψουμε το πράσινο φως, δεν θα ήταν κακό το Ευρωκοινοβούλιο να δίνει κάποια κατεύθυνση διαδικασία. Δεν είναι πολύ δημοκρατικό στο τέλος να αντιμετωπίσουμε ένα τελικό αποτέλεσμα χωρίς να έχουμε τη δυνατότητα κάπως να διαμορφώσουμε αυτό το αποτέλεσμα. Δεν έχουμε κάποιες ενδείξεις τώρα για ύπαρξη άλλων εγγράφων περιμένουμε. Ελπίζουμε να τα παραλάβουμε τις επόμενες ημέρες. Έγγραφα που θα αφορούν τα διάφορα ζητήματα. Τι είπατε? Όχι. Ελπίζω για μέρες μόνο να περιμένουμε. Όχι για χρόνια. Σίγουρα. Όπως έχουμε αναφέρει στην πρόσφατη θέση μας που εκφράσαμε αν κάποιο αναφέρει ότι πρέπει να επιτευχθεί επαρκή πρόοδος γιατί να μπούμε στη δεύτερη φάση των διαπραγματεύσεων, επαρκή πρόοδος τι σημαίνει. Ότι σε ένα τομέα έχουν επιτευχθεί, ε, έχει επιτευχθεί πρόοδος και όχι σε, άλλη, σε άλλο τομέα. Αυτό δεν είναι πρόοδος για μένα. Πρέπει όλοι οι τομείς να προχωρούν. Να σημαίνονται πρόοδος σε όλου του τομεί. Δεν μπορεί να προχωράει ένα κομμάτι των διαπραγματεύσεων και στα υπόλοιπα θέματα να μην έχουν προχωρήσει αρκετά. Επαρκής πρόοδος, επαρκές τι σημαίνει. Όπως και στην ομάδα το αναφέραμε τον Brexit, ότι σε όλα τα θέματα σημειώνεται πρόοδος. Οπότε έτσι έρχομαι σε αυτό που είπε και ο Σόλτς, που αναφέρθηκε σε προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών εγώ είμαι ένθερμος υποστηρικτής της ταχύτερης ε, βεβαιότητας που θα δοθεί στους πολίτες και στους πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου και τους πολίτες Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί. Υπό μια προϋπόθεση βέβαια. Να αναγνωρίσει το Ηνωμένο Βασίλειο το ταχύτερο δυνατόν ότι χρειάζεται κάποια οικονομική διευθέτηση. Δεν λέω ότι χρειαζόμαστε συμφωνία τώρα ήδη όσον αφορά τα αριθμητικά στοιχεία τα συγκεκριμένα. Αυτό ε, είναι δύσκολο για πολιτική διαπραγμάτευση. Να υπάρξει συμφωνία επί της αρχής. Αυτό θα βοηθούσε. Αυτή η αναγνώριση από το Ηνωμένο Βασίλειο ότι υπάρχει ανάγκη οικονομικής διευθέτησης θα βοηθούσε την επιτάχυνση και των άλλων σημαντικών διαπραγματεύσεων για τα άλλα σημαντικά ζητήματα και κυρίως για το θέμα των δικαιωμάτων των πολιτών. Υπήρξε και άλλο ερώτημα για, τον, για το Horizon 2020 και για το Εράσμου σε συμφωνία σύνδεσης βάσει του άρθρου 2.17 όλα αυτά τα προβλήματα αντιμετωπίζονται. Διάφορες χώρες συμμετείχαν στον ορίζοντα 2020 χωρίς να είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Το Ισραήλ είναι ένα τυπικό παράδειγμα αυτού. Αλλά αυτό συνεπάγεται δικαιώματα αλλά και υποχρεώσεις. Πληρώνουν γι' αυτό. Κανονικό είναι αυτό στον ορίζοντα 2020 στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Από όλες τις πλευρές δεν υπάρχει πρόβλημα εμπόδιο να βρεθούν τρόποι συνεργασίας στο έρασμος, στον ορίζοντα 2020 και σε άλλους τομείς. Αλλά δεν θα είναι δωρεάν. Δεν είναι δωρεάν γεύμα, δεν υπάρχει αυτό. Ίσως κάποιοι να διατείνονται ότι υπάρχει. Αλλά ο απλός άνθρωπος θεωρεί ότι κανονικά πρέπει να πληρώσει για το γεύμα του. Τέλος, θα απηχήσω τα υποθέντα από την Πρόεδρο. Εδώ δεν τίθεται θέμα αριθμών. Τρία εκατομμύρια από εδώ έχουμε πολίτες και ένα εκατομμύριο από την άλλη, αυτό που αναφέρατε. Και εγώ θα, θα μπορούσα... Ε, είναι 0,6% του συνολικού πληθυσμού τα 3 εκατομμύρια και το 1 εκατομμύριο Βρετανών που έχονται στην Ήπειρο ότι προσωπεύει περίπου 2% του συνολικού βρετανικού πληθυσμού. Τι νόημα έχουν αυτά τα νούμερα. Μιλάμε για πολίτες, μιλάμε για ανθρώπους, για άτομα. Κάθε άνθρωπος, ακόμα και αν μιλάμε για ένα άτομο και μόνο, μία μόνο οικογένεια, πρέπει να μεριμνήσουμε γι' αυτό. Δεν είναι θέμα αριθμών. Είναι θέμα ανθρωπίνων όντων. Δεν μπορείς να εκφράζεσαι με αριθμού για αυτά τα θέματα. Αμοιβαιότητα είναι αμοιβαιότητα στα δικαιώματα δεν μπορεί να πει κανεί ότι έχουμε μόνο εκατομμύριο εδώ και τρία εκατομμύρια εκεί συμφέροντα. Μιλάμε για ανθρώπου. Για την άποψή μου. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Και το συνέστημά μου δεν μπορεί να κινηθεί σε αυτά τα θέματα με αριθμού. Σκεφτείτε και κάτι άλλο. Οι υπήκοοι του Ηνωμένου Βασιλείου που εργάζονται στην Ήπειρο φέρνουν και δίνουν κάτι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και οι πολίτες που ζουν στην Βρετανία και αυτοί συνεισφέρουν στην ευημερία και στην οικονομία της Βρετανίας. Ας τα δούμε θετικά και όχι σαν βάρος. Οι άνθρωποι δεν είναι βάρος. Και οι άνθρωποι είναι στο επίκεντρο των δράσεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. ευχαριστώ. Καταφέραμε να τηρήσουμε το χρόνο. Κύριε Πρέσβη, ε, φτάσατε ακριβώς στην κατάλληλη στιγμή. Ευχαριστώ πολύ να κλείσουμε αυτό το θέμα και περνάμε στο τελευταίο θέμα στη μέση διάταξη <clears throat> που είναι ο απολογισμός της ε, Μαλτέζικης Προεδρίας. Σας παρακαλώ, πρέπει να φύγουν, να φύγουν, να αποχωρήσουν ησυχώς. Συνεχίζεται η συνεδρίασή μας. Να καλωσορίσω από πλευρά σας την κυρία Μαρλίν Μπονίτσι από τη Μάλτα. Μαλτέζικη Προεδρία κατέληξε. Ακόμη και τα πιο θαυμάσια πράγματα κάποια στιγμή τελειώνουν. Θα ήθελα λοιπόν να μας κάνετε τον απολογισμό της Προεδρίας σας. Οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Εσείς θα επιλέξετε τα θέματα και έχετε όσο χρόνο θέλετε. Παρακαλώ. Uh, Ευχαριστώ κυρία Χούμπνερ. Με χαρά είμαι εδώ για να σα παρουσιάσω τα θέματα που αντιμετώπισε η Μαλτέσκη Πρεδρία. Ο Υπουργός μου θα ήθελε πολύ να είναι εδώ αλλά όπως θα ξέρετε όσοι παρακολουθείτε την ε, πολιτική κατάσταση στην Μάλτα θα ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή συζητάει ένα κρίσιμο νομοθέτημα στο κοινοβούλιο μας που ελπίζουμε να εγκριθεί σήμερα. Τώρα η Προεδρία μας. Τι επέτυχε. Συνέχισε να εργάζεται σε μια σειρά από βασικά θέματα που ενδιαφέρουν ιδιαίτερα την Επιτροπή σας συμπεριλαμβανομένη της τροποποίησης του εκλογικού νόμου και το μητρό διαφάνειας. Αλλά με περιορισμένη επιτυχία. Ξέρουμε πόσο περίπλοκα είναι τα θέματα αυτά. Και λεπτά. Για την τροποποίηση του εκλογικού νόμου. Παρά τη σκληρή δουλειά που έκανε η Τρόικα προεδριών, η Ολλανδική, η Μαλτέζικη και η Εστονική, δεν επέδευξαν πολλά. Και το αυτό ισχύει και για το Μητρό Διαφάνειας. Συνεχίζεται η εργασία. Κατά την Προεδρία μας επιτύχαμε τουλάχιστον συμφωνία να γίνει η πρώτη τριμερή συνάντηση σε πολιτικό επίπεδο, αλλά λόγω των υποχρεώσεων των συμμετεχόντων δεν ε, συμφωνήθηκε η ημερομηνία. Για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα, για το καθεστώς τους, ε, χαιρετίζουμε την αρχή ισχύω ε, του νέου κανονισμού και κατά την Προεδρία μας επιτύχαμε να ορίσει το Συμβούλιο τους δύο εκπροσώπους του για την εφαρμογή των, του, II, α, του της Διοργανικής Συμφωνίας. Νομίζω ότι επετεύχθη αρκετή πρόοδος για τις διεθνείς συμφωνίες είχαμε πολλές συζητήσεις σε τεχνικό επίπεδο έγινε μια προσπάθεια καθορισμού του πεδίου εφαρμογής και καταλήξαμε στην πολιτική συνάντηση της 4ης Ιουλίου προσπαθήσαμε να λάβει χώρα κατά την Προεδρία μας αλλά και πάλι υποχρεώσεις των συμμετεχόντων δεν το επέτρεψαν αλλά σημειώνω με ικανοποίηση ότι τελικά διεξήχθη την 4η Ιούλιου και από ό,τι έμαθα πήγε πολύ καλά όλα τα θεσμικά όργανα συμφώνησαν ε, σε μια επικοδομητική προσέγγιση για τις μελέτες αντικτύπου. Η Προεδρία μας πρώτα απ' όλα κατάφερε να καταλήξει σε μια προσέγγιση για το θέμα αυτό για τις περιπτώσεις ε, στις οποίες χρειάζεται. Υπάρχει διαδικασία καθορισμού τους για τις ε, κατεξοδότηση και εφαρμοστικές πράξεις. Το Συμβούλιο ξεκίνησε να μελετάει την πρόταση της Επιτροπής. Όλοι ξέρουμε ότι ε, ιδιαίτερα μακροσκελής Επιτεύχει μεγάλη πρόοδο για διάφορους τομείς της πρότασης. Η Μαλτέζικη Προεδρία κάλυψε 10 από τα 13 τμήματα του κειμένου της πρότασης Επιτροπής. Και κάναμε απολογισμό της προόδου σε μια έκθεση προόδου την οποία υπέβαλε στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων 28 Ιουνίου η Μαλτέζικη Προεδρία. για το καθορισμό των μη δεσμευτικών κριτηρίων για την εφαρμογή του 290 και 291 της συνθήκης, στο Συμβούλιο επανήλθε στο Κοινοβούλιο εκφράζοντας την βούλησή του να ε, υπάρξει έναρξη των διαπραγματεύσεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή. Και παράλληλα. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρξει πρόοδος στο θέμα ευθυγράμμιση πρακ. Ελπίζουμε να συνεχιστεί αυτή η συζήτηση και κατά την επόμενη Προεδρία, δηλαδή την παρούσα. Για την εφαρμογή της κοινή ε, δήλωσης υπήρξε μια συζήτηση σε πολιτικό επίπεδο μεταξύ της Προεδρίας του, του Συμβουλίου και της Προέδρου Σταγιάννη και Γιούνκερ Συζητήσαμε την πρόοδο σε συγκεκριμένα θέματα που περιέχονταν στην κοινή δήλωση και η προσπάθεια αυτή έδειξε τη σημασία της συνεργασίας των τριών θεσμικών οργάνων. Το Συμβούλιο άρχισε την εργασία του για το πρόγραμμα εργασίας για το 2018 και κάναμε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων του παρελθόντος Ιουνίου. Για τον Brexit, ε, ξέρω ότι μόλις το συζητήσατε, αλλά να σας πω τι έκανε η Προεδρία μας. Μετά την ε, ενεργοποίηση του άρθρου 50, ό,τι δηλαδή προτίθεται το Βασίλειο να αποχωρήσει από, το, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά λοιπόν αυτή την κοινοποίηση 29 Μαρτίου το Συμβούλιο εργάστηκε ταχύτατα και τον Απρίλιο υιοθετήθηκαν οι χαρακτηριστικές γραμμές από το Συμβούλιο Κορυφής και το Μάιο εγκρίθηκαν οι διαπραγματευτικές οδηγίες στις 29 Μαΐου. Και χαιρετίζουμε και τη Συμβουλή την συμβολή του Κοινοβουλίου σε αυτή τη διαδικασία και ήμασταν καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας και της Προεδρίας μας σε επαφή με το Κοινοβούλιο. Υπήρξε ανταλλαγή απόψεων και πριν και μετά το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων μεταξύ του Προέδρου του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων και του εκπροσώπου σας για θέματα Brexit. Ο χρόνος πιέζει, η ταχεία έγκριση των οδηγιών σήμαινε ότι ήμασταν σε θέση να ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις αμέσως μετά τις εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες τώρα έχουν ξεκινήσει. Προτεραιότητα δίδεται στα δικαιώματα των πολιτών, την οικονομική διευθέτηση και τα συνοριακά θέματα. Το Μάιο και τον Ιούνιο το Συμβούλιο έδειξε την αποφασιστικότητά του ότι θέλει να δράσει ούτως ώστε το Brexit να δημιουργήσει τα λιγότερα προβλήματα στη λειτουργία της Ένωσης, τις λιγότερες διαταραχές. Επίσης, εργαζόμεθα και στο θέμα της μετεκατάστασης των δύο φορέων που είναι στο Λονδίνο, τον, ε, του Οργανισμού Φαρμάκων και της Αρχής για τις Τράπεζες. Εργαστήκαμε μια σειρά από εβδομάδες και οι αποφάσεις ε, υιοθετήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και προβλέπουν ότι η τελική απόφαση για τη μετακατάσταση των δύο οργανισμών θα ληφθεί το προσεχές φθινόπωρο. Φυσικά το να καθορίσουμε το θέμα των οργανισμών πολύ νωρίς θα μας διασφαλίσει να μπορούν να λειτουργούν σε άλλη έδρα αυτοί οι δύο οργανισμοί πριν την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου που είναι ουσιώδες για να υπάρχει συνέχεια στις ουσιώδες υπηρεσίες που παρέχουν και οι δύο αυτοί οργανισμοί για την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ένταξη δηλαδή της Ένωσης ε, σε αυτήν, προγραμματίσαμε μια σειρά από συναντήσεις, αλλά υπήρξε και η απόφαση τέλη Μαρτίου τρέχοντος και το Συμβούλιο έκτοτε περιμένει η Επιτροπή να δώσει την τεχνική της σύμβολη. Αυτή είναι μια γενική επισκόπηση της εργασίας που επετέλεσε η Προεδρία μας και για πολλά από αυτά τα θέματα είμαι πεπισμένη ότι θα υπάρξουν περαιτέρω εξελίξεις υπό την παρούσα. Προεδρία, ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Τζόρτς Σέπλιν έχει το λόγο. Ευχαριστώ και την κυρία Πρέσβη και την Πρόεδρο. Σα ευχαριστώ ιδιαίτερα κυρία μου που ήρθατε εδώ για να μα παρουσιάσετε τι κάνατε τις, ε, τους τελευταίους έξι μήνε. Ε, ξέρω πόσο δύσκολη είναι η πρώτη προεδρία. Θυμάμαι τι είχε γίνει με την Ουγγαρία στην αντίστοιχη θέση. Θέσατε κάποια θέματα και θα ήθελα να σταθώ εκεί. Είπατε πως για τον εκλογικό νόμο ήταν περιορισμένη η πρόοδος. Μήπως μπορείτε να μας περιγράψετε τα εμπόδια τα οποία αντιμετωπίσατε, κάποια τα οποία ίσως ξεπεράσατε. Ε, πού ακριβώς είναι η κατάσταση σήμερα και για τα πολιτικά κόμματα. Και πάλι αναφερθήκατε στην ε, αρχική σας παρουσίαση στο θέμα αυτό και θα ήθελα να μου πείτε πού έχουμε φτάσει. Τέλος, έχω μια τεχνική ερώτηση για το Brexit. Πόσοι Μαλτέζοι επηρεάζονται από το θέμα αυτό, γιατί ξέρετε πως ε, αν δεν κάνω λάθος, ψήφισαν στο δημοψήφισμα γιατί ανήκουν στο Commonwealth, αλλά πείτε μου, με υπηκότητα Μάλτας, πόσοι είναι οι άνθρωποι που ζουν στην ε, Βρετανία. Κοιτάξτε, τους μετρήσαμε, αλλά όσο μετράμε τόσο αυγατίζουν, γιατί ξέρετε πως πολλοί ζουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια στο Ηνωμένο Βασίλειο με τη δική μας υπηκότητα και μετά την ένταξη ε, της Μάλτας στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι περισσότεροι δεν ζήτησαν τη δική μας υπηκότητα γιατί όσοι έχουν δικαίωμα να την ε, ζητήσουν, να την αιτηθούν. Για παράδειγμα, τα παιδιά της πρώτης γενιάς των Μαλτέζων που μετακινήθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν έκανα κάτι τέτοιο. Λόγω Brexit όμως, πολλοί από αυτούς που έχουν το δικαίωμα ε, βρίσκονται στη διαδικασία αίτησης. Οπότε ελπίζω να δούμε σύντομα τι γίνεται. Εμείς κοιτάξαμε τα στοιχεία στο Υπουργείο Εξωτερικών και μας είπαν πως είναι ένας αριθμός ε, που αλλάζει σχεδόν σε καθημερινή βάση. Για τα υπόλοιπα δύο να σας πω πως σε γενικές γραμμές τα θέματα τα οποία αντιμετώπισε η Προεδρία μας ήταν αυτά τα οποία αντιμετώπισαν και οι προηγούμενοι δεν έχουμε κάτι το καινούριο να σας παρουσιάσουμε. Ξέρετε πως έχουν γίνει αρκετές συζητήσεις και τρέχουν εδώ και περίπου 1,5 χρόνο για τα διάφορα θέματα. Έχουμε μία πρώτη συμφωνία σε ελάχιστα μόνα σε ελάχιστες μόνες, μόνο τροποποιήσεις, ε, οι οποίες είναι περισσότερο ε, συμβολικού χαρακτήρα, ψηφοφορία μέσω διαδικτύου, ανταλλαγή πληροφοριών, έτσι ώστε τα κράτη-μέλη να μπορέσουν να αποφασίσουν ε, πόση ορατότητα θα δώσουν στα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και πώς αυτό θα εμφανίζεται με γραφικά πάνω στα ψηφοδέλτια. δεν έχω κάποια απτά αποτελέσματα να σας παρουσιάσω. Και το ίδιο ισχύει και για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα. Το βασικό μήνυμα από τη δική μας πλευρά ήταν πως καταφέραμε το Συμβούλιο να συμφωνήσει ποιοι θα είναι οι δύο εκπρόσωποι του και δεν νομίζω ότι καταφέραμε να κάνουμε πολλά παραπάνω από αυτό. Δεν γνωρίζουμε πώς θα προχωρήσει το θέμα αυτό και αν σημειωθεί μεγαλύτερη πρόοδος, πίσω το Συμβούλιο θα μπορούσε να εξετάσει και τροποποίηση του κανονισμού του 14. Δυστυχώς όμως κατά τη δική μας Προεδρία και λόγω των ίδιων λόγων και ζητημάτων που έχουν επηρεάσει άλλες Προεδρίες, παρόλες τις πολλές προσπάθειες που κάναμε, δεν στάθηκε δυνατό. και τα ίδια θέματα ε, εξακολουθούν να προκύπτουν ε, όταν τα συζητάμε στο Συμβούλιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Να σας πω μόνο πως ε, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για την πολύ λεπτομερή ενημέρωση που μας κάνατε και ελπίζω πως η πρώτη πολιτική συνάντηση για τη διαφάνεια θα γίνει. Δεν μπορέσαμε να το κάνουμε παρουσία σας. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουμε και με τους εστονούς. Εν πάση περιπτώσει θα προσπαθήσουμε μετά ε, το καλοκαίρι. Σας ευχαριστώ και για την έκθεσή σας για το Brexit. Συνήθως μιλάμε με τον Μισελ Μπαρνιέ, με εκπροσώπους Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οπότε νομίζω πως είστε η πρώτη προεδρία η οποία μοιράζεται μαζί μας τα θέματα αυτά. Και ίσως γιατί αυτή τη στιγμή ε, έχουν προκύψει περισσότερα από ό,τι ε, πριν από εσά σε άλλε προεδρίε. Τώρα, για την προσχώρηση στη σύμβαση για, την, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ξέρω πω για κάποιου συναδέλφου τώρα που βρίσκονται εδώ είναι σημαντικό. Μα είπατε μετά την απόφαση του Μαρτίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σα έχει υποσχεθεί να καταθέσει κάποιο έγγραφο. Μπορείτε να μα δώσετε κάποιε λεπτομέρειε. Οι πληροφορίε που έχω είναι πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καταθέσει τεχνικές συνεισφορές Ο στόχος μας ήταν να προχωρήσουμε αφού κατατεθούν αυτές οι τεχνικές λεπτομέρειες προς συζήτηση στο Συμβούλιο. Αλλά δυστυχώς δεν τις λάβαμε και από ό,τι με ενημερώνουν και υπό την πρώτη, υπό, κατά την πρώτη υποστονική προεδρία συνάντηση δεν ε, έφτασαν αυτές οι τεχνικές ε, συνεισφορές. Καταλαβαίνω βέβαια πως είναι ε, τεχνικά και νομοτεχνικά ζητήματα, αλλά η σχετική ομάδα εργασίας υπό τη δική μας προεδρία ήταν έτοιμη για να τα εξετάσει. Παρ' όλα αυτά δεν μπορέσαμε να κάνουμε και πολλά, γιατί επαναλαμβάνω ε, έλειπαν τα έγγραφα με τις τεχνικές λεπτομέρειες από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ξέρω πως κάθε, κάποιοι συνάδελφοι από την Κομισιόν κάθονται ε, ε, εκεί πίσω, οπότε σας παρακαλώ πολύ να μεταφέρετε το μήνυμα αυτό από το Ευρωκοινοβούλιο και από το Συμβούλιο. Περιμένουμε. Περιμένουμε τα κείμενα ε, με τις τεχνικές προτάσεις. Θα ήθελα να το επαναλάβετε. Αν δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, δεν ξέρω, ο Τζόρτζ, έχει τελειώσει, ο Χέλ μου την εντάξει. Μία ερώτηση, σύντομη, αφού σας ευχαριστήσω για τα όσα έχετε κάνει, για τις διεθνείς συμφωνίες. Είπατε πως γίνεται αυτή τη στιγμή επικοδομητική προσπάθεια πρόοδου. Τι ακριβώς εννοείτε όταν λέτε επικοδομητικό, τι ακριβώς εννοείτε, ποια είναι τα προβλήματα και τι θα έπρεπε να συζητήσουμε και μεταξύ μας για το τι μπορούμε να κάνουμε από την πλευρά του Κοινοβουλίου. Και πάλι δεν ήμουνα στις 4 Ιουλίου γιατί είχε λήξει πια η Προεδρία μου αλλά μπορώ να σας πω πως κατά τη δική μας Προεδρία προσπαθήσαμε να κάνουμε τις αφανείς εργασίες σε τεχνικό επίπεδο γνωρίζοντας ποιες είναι οι προσδοκίες του Κοινοβουλίου και μέχρι πού μπορεί να φτάσει στο Συμβούλιο. Επίσης κάναμε και κάποιες άτυπες συζητήσεις με το Συμβούλιο για να προσπαθήσουμε κάθε φορά να επιστρέψουμε με κάποιο είδους πρόοδο. Επαναλαμβάνω, στις 4 Ιουλίου στη συνάντηση δεν ήμουν, αλλά μίλησα με κάποιους οι οποίοι με ενημερώνουν πως έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος, τουλάχιστον σε σχέση με τις προσδοκίες του Κοινοβουλίου, και πως έχει σημαντηθεί επίσης μεγάλη πρόοδος στο θέμα της δέσμευσης του Συμβουλίου. Ακόμα βέβαια το Συμβούλιο δεν είναι σε θέση να συμφωνήσει πλήρως για όλα τα θέματα. Ξέρετε εξίσου καλά με εμένα που τα δύο ζητήματα είναι πρώτον τα κριτήρια στα πλαίσια των διαπραγματευτικών οδηγιών και η προσωρινή εφαρμογή των συμφωνιών. Και ενημερώνομαι πως τα αποτελέσματα της συνάντησης αυτής θα μεταφερθούν στο Συμβούλιο για να εκφράσει την άποψή του, αλλά ήταν εξαιρετικά επικοδομητική η συνάντηση και από όλες τις πλευρές και για την προσωρινή εφαρμογή και εκεί ακόμα η υπηρεσία εξαιρετικής δράσης είπε ότι θα κοιτάξει την ε, συνθήκη και θα δει τι μπορεί να κάνει. Λυπηθήκαμε βέβαια που αυτό δεν μπορούσε να γίνει που τη δική μας Προεδρία. Είχαμε προετοιμαστεί πάρα πολύ γερά, αλλά βέβαια υπήρχαν θέματα χρονικού προγραμματισμού και αυτό πάντα συμβαίνει ότι αν φτάνει κανείς προς το τέλος Προεδρίας του, δηλαδή ξαφνικά αρχίζει να μην έχει χρόνο. Πάντως είμαι ικανοποιημένη που στο Συμβούλιο από τη μία Προεδρία ε, στην επόμενη δουλεύουμε καλά και πραγματικά η ενημέρωση που έλαβα ήταν πως ο χρόνος που διαθέσαμε εμείς στην προετοιμασία αυτών των συναντήσεων τελικά ε, χρησιμεύσε. Ευχαριστώ πολύ να προσθέσω γιατί ακούσαμε τον Λάγκη και τον Μπρόκ στην σχετική συνάντηση και υπάρχει ένα θέμα το οποίο δεν έχει συμφωνηθεί στο Συμβούλιο που ήταν η προσωρινή εφαρμογή, ο ρόλος του Κοινοβουλίου και χαίρομαι που το αναφέρατε κι εσείς αλλά θα καλέσουμε τους συναδέλφους να μας υποβάλουν τη σχετική έκθεση. λοιπόν, δεν υπάρχουν άλλα σχόλια. Σας ευχαριστώ. Σας συγχαίρω. Θα χαρήκατε κι εσείς που μπορείτε να χαλαρώσετε. Ξέρω πως οι πρέσβεις πάντα για έξι μήνες είναι στη χειρότερη θέση. Σας ευχαριστώ και ελπίζω πως θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τη Μάλτα. Αν όχι βέβαια ως Προεδρία, αλλά ως ε, μεμονωμένο κράτος μέλους. Συνάδελφοι. Η πρωινή μας συνεδρία λίγη θα τα ξαναπούμε στις 3. Οπότε, στις 3 για να συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα.